Bien, συνάδελφοι, καλώ ήρθατε. Να σα πληροφορήσω ότι υπάρχει μια αλλαγή προγράμματο για σήμερα το απόγευμα. Δυστυχώ, δεν μπορούμε να κάνουμε τη συνάντηση που προβλεπόταν με τον κύριο Άλεξ Ρόντο, τον ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κέρας της Αφρικής διότι χρειάστηκε να ξαναφύγει κατεπηγώντας χθε για διαπραγματεύσει μεταξύ του Σουδάν και του Βορείου του Νοτιού Σουδάν. Δεν θα είναι δυνατό λοιπόν να έχουμε αυτό το τμήμα της συνεδρίασής μας στο απόγευμα. Και επειδή δεν έχουμε πραγματικά χρόνο, μάλλον επειδή μας πληροφορήσαν τελευταία στιγμή, δεν μπορέσαμε να οργανώσουμε μια εναλλακτική συνεδρίαση το απόγευμα για άλλα θέματα. Υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία όμως δεν βρίσκονται στις προτεραιότητες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Προτιμώ λοιπόν να μην κάνουμε καθόλου συνεδρία στο απόγευμα παρά μια συνεδρίαση η οποία θα, δεν θα έχει ουσιαστικό περιεχόμενο. Επομένως θα συνεδριάσουμε το απόγευμα. Σήμερα όμως έχουμε αρκετά σημεία στην μέση για διάταξη. Καταρχήν την πολιτική αποστολή για το Μαλί, η οποία είναι σε επίπεδο προγραμματισμού. Επίσης τη στρατηγική ασφάλεια για την ασφάλεια στη θάλασσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι από τις σπάνιες φιλόδοξες ανακοίνωσης του Συμβουλίου κορυφής του Δεκεμβρίου και επίσης έχουμε την Ευρωπαϊκή Διοίκηση Ευρωμεταφορών και αυτό είναι μια από τις σπάνιες επιτυχίες στην θέση από κοινού των πόρων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινάμε λοιπόν με το Μαλί. Χαιρετίζω τον Didier Lenoir, ο οποίος ασκεί χρέη διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κρίσεων και Σχεδιασμού της AEF. Στις 17 ε, Μαρτίου στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών συζητήθηκε η ανάπτυξη μιας πολιτικής αποστολής ε, στο Μαλί, διότι υπάρχει ήδη μια στρατιωτική αποστολή όπως γνωρίζετε εδώ και ένα χρόνο, η οποία λειτουργεί πολύ καλά και ο Διδιά ίσως μπορεί να πει κάτι σχετικά, αλλά λειτουργεί με ικανοποιητικό τρόπο αυτή η αποστολή. Περιλαμβάνει <clears throat> συνεισφορές από διάφορες ε, χώρες 23, αν δεν κάνω λάθος. Επομένως είναι μια πραγματική επιτυχία και τώρα ο στόχος της προετοιμαζόμενης πολιτικής αποστολής είναι η κατάρτιση των δυνάμεων ασφαλείας στο Μαλί και ο Ντιδία θα επανέλθει στο θέμα αυτό για το υπόδειγμα αυτό που θα ακολουθηθεί το οποίο χρησιμοποιήθηκε ήδη στην περίπτωση του Νίγηρα, μιας γειτονική χώρας και είναι ενδιαφέρον να δούμε σε ποιο πλαίσιο μπορεί να εγγραφεί αυτή η αποστολή, πώς θα αλληλεπιδράσει με τη στρατιωτική αποστολή, πώς θα ε, συνδυαστεί με την πολιτική αποστολή που βρίσκεται σε μια γειτονική χώρα των ε, Νίγηρα, αν μπορεί να δημιουργηθεί μια πολιτική αποστολή περιφερειακού χαρακτήρα για όλες τις χώρες της περιοχής, ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα, ποιος είναι ο αριθμός των ε, ατόμων των ανδρών που θα αναπτυχθούν. Θα ήταν πολύ χρήσιμο λοιπόν να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες για αυτή την αποστολή. Και νομίζω το καλύτερο είναι να σας δώσω το λόγο να μας παρουσιάσετε την κατάσταση των πραγμάτων στην Ε.Ε. και μετά μπορούμε να συνεχίσουμε με μια ανταλλαγή ερωτήσεων και απαντήσεων. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας πληροφορήσω για, τα, για τις εργασίες Παρασκευής της πολιτικής αυτής αποστολής. Έχει κρατήσει αρκετό καιρό η εκόλαψη ούτως υπήν αυτής της αποστολής. Ξεκίνησαν συζητήσεις τον Ιούλιο του 2013 αλλά μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα μπορέσαμε να διαμορφώσουμε καλύτερα ένα λειτουργικό, <clears throat> ένα επιχειρησιακό μάλλον και στρατηγικό πλαίσιο για αυτή την αποστολή στο Μαλί και νομίζουμε τώρα ότι έχουμε μια πράγματι σταθερή βάση για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε αυτή την πολιτική αποστολή. Ο στόχος αυτής της αποστολής δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται ως έκπληξη, είναι κάτι το οποίο εγγράφεται πλήρως στη λογική της στρατηγικής για, τις περιοχές, για, τη χώρα του, για τις χώρες του Σαχέλ που ενεκρίθη από το Συμβούλιο και επίσης συνδέεται με την ε, χρηματοδοτική βοήθεια που δόθηκε στο Μαλί. 615 εκατομμύρια για τα επόμενα χρόνια από το Περιφερειακό Ταμείο και επίσης συνδέεται με την ε, δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, στρατιωτική συνεργασία με την κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας και τη στρατιωτική αποστολή. Όταν ξεκινήσαμε τη στρατιωτική αποστολή Είχαμε πει σαφώς ότι αυτή η στρατηγική αποστολή για να μπορέσει να επιτύχει τους πολιτικούς στόχους που επιζητούσε θα πρέπει να, να συνοδεύεται από μια πολιτική αποστολή. Σας υπενθυμίζω ότι εμείς ήμασταν στο Μαλί, ήρθαμε στο Μαλί εξ ονόματος της ΚΕΠΑ, διότι υπήρχε απόλυτη έλλειψη κράτους δικαίου και κρατικού ελέγχου στο Βόρειο Μαλί. Αυτό ήταν μια πηγή απειλών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Μαλί ήταν ένας χώρος λαθρεμπορίων, τρομοκρατίας, που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο και επομένως ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν να επιτρέψει το κράτος του Μαλί να αναλάβει και πάλι τον έλεγχο του Βορείου Μαλί... για να αποφύγει να είναι το Βόρειο Μαλί ένας χώρος για την ανάπτυξη απειλών για την εσωτερική ασφάλεια του Μαλί και ευρύτερα. Αν σκεφτούμε λοιπόν αυτό το στόχο καταλαβαίνουμε πολύ γρήγορα ότι οι καλύτερες δυνάμεις και οι πιο εύστοχες για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε της, ε, την ασφάλεια του βόρειου τμήματος του Μαλή θα ήταν οι εθνικές δυνάμεις ασφαλείας. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με τη στρατιωτική αποστολή για να μπορέσουν να αναπτυχθούν αυτές οι δυνάμεις σε ένα ασφαλές πλαίσιο και αυτό ήταν το τμήμα το οποίο αφορούσε το στρατό του Μαλή. Με τη δική μας παρουσία μπόρεσε ο στρατός του Μαλή να ελέγξει καλύτερα το βόρειο τμήμα του, <clears throat> του Μαλή ώστε οι δυνάμεις της τάξης, η αστυνομία, οι δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας μπορούν να, να μπορέσουν να εξασφαλίσουν το κράτος δικαίου και την ασφάλεια στην περιοχή αυτή. Και αυτή ήταν η βασική σκέψη που οδήγησε στην εκκίνηση αυτής της στρατιωτικής ε, ε αποστολής. Δεν έγινε η αποστολή μόνο και μόνο για να γίνει. <clears throat> και αυτή ήταν η βασική οδηγός γραμμή από την αρχή της παρουσίας μας στο Μαλί. Τώρα, πρόσφατα το Συμβούλιο ενέκρινε την ιδέα του να υποστηριχθούν οι αρχές του Μαλί στη μεταρρύθμιση που πρέπει να κάνουν στο, στις δυνάμεις ασφαλείας τους. Πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και βελτίωση του έργου των δυνάμεων ασφαλείας στο εσωτερικό. Καταρχήν μας ενδιαφέρει να ευνοήσουμε και να ενισχύσουμε την επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων αυτών. Πρόκειται για μια αποστολή κατάρτισης λοιπόν. Δεύτερον, να υπάρχει καλύτερη στελέχωση και διοίκηση αυτών των δυνάμεων. Επομένως, πρόκειται για εργασία σε σχέση με τα ανώτερα στελέχη. Τρίτον, θα πρέπει αυτά τα ανώτερα στελέχη να ελέγχονται από την πολιτική εξουσία και να συνεργάζονται με τις δικαστικές αρχές γιατί υπήρξε ένα πρόβλημα <clears throat> σύνδεσης μεταξύ αστυνομία και δικαιοσύνης. Επομένως ο στόχος θα πρέπει να είναι να βελτιώσουμε τον έλεγχο από τις διοικητικές αρχές στις ε, αστυνομικές και άλλες δυνάμεις ασφαλείας. Τέταρτον, από τη στιγμή που θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτό το συνεκτικό πλαίσιο και που ελπίζουμε θα είναι πιο αποτελεσματικό, να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη αυτών των δυνάμεων στο βόρειο τμήμα του Μαλή και να υποστηρίξουμε σε επίπεδο επιμελητίας και οργάνωσης αυτή την ανάπτυξη. Επομένως, το χρονοδιάγραμμα ε, είναι ότι μόλις έχει εγκριθεί η βασική αρχή για αυτή την αποστολή, το πρώτο στάδιο είναι τώρα να οργανωθεί αυτή η αποστολή, η πολιτικού χαρακτήρα αποστολή, κάτι το οποίο θα γίνει πολύ γρήγορα. Αυτό προβλέπεται να ξεκινήσει τα, στα μέσα Απριλίου με μια σημαντική ομάδα που θα περιλαμβάνει και τον επικεφαλή τη αποστολή. Η ομάδα αυτή θα ε, κάνει την εγκατάσταση της αποστολής, θα δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές και δίκτυα και στη συνέχεια θα εργαστεί για να αναπτύξει ένα επιχειρησιακό σχέδιο σε στενή συνεργασία με τις αρχές του Μαλή. Η ελπίδα μας λοιπόν είναι ότι θα μπορέσουν να προχωρήσουν αυτά πολύ γρήγορα και το επόμενο στάδιο θα είναι η πλήρης ανάπτυξη αυτής της αποστολής. ελπίσουμε ότι σε λίγους μήνες, σίγουρα πριν από το τέλος του 2014, αυτή η αποστολή θα είναι πλήρως λειτουργική, θα έχει γίνει ο σχεδιασμός, θα έχει αναπτυχθεί και θα είναι σε θέση να αρχίσει τις δραστηριότητές της. Για να επιταχύνουμε κάπως το χρονοδιάγραμμα αυτό, χρησιμοποίησαμε κάποιες νέες διαδικασίες. Ξέρω το θέμα της ανάπτυξης πολιτικών αποστόλων είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί πολλές φορές. Και εδώ Υπάρχουν νέε διαδικασίε, προσπαθήσαμε μαζί με του συναδέλφους μα οι οποίοι ελέγχουν το, τη σχεδίαση των αποστολών να κάνουμε τη λεγόμενη παράλληλη σχεδίαση, δηλαδή να εξασφαλίσουμε ότι η στρατηγική σχεδίαση μετά από τι αποφάσει του Συμβουλίου τη 17 7η Μαρτίου να γίνεται παράλληλα με την επιχειρησιακή <clears throat> σχεδίαση ώστε να μπορούμε από τι πρώτε εβδομάδε να αναπτύξουμε κάποιε ομάδε. Για τους πόρους τώρα αυτής της ε, αποστολής. Δεν έχει ακόμα καθοριστεί ο αριθμό των ατόμων που θα λάβουν ε, μέρο. Αυτό θα, χαρα... θα καθοριστεί μέσα στην επιχειρησιακή σχεδίαση. Αλλά εκτός εκπλήξεων θα είναι ανάλογο το μέγεθος αυτής της αποστολής με την αποστολή στον Ήγηρα. και τίθεται επίση και το θέμα των πόρων που θα πρέπει να δοθούν σε αυτήν την ε, αποστολή, η οποία χρηματοδοτείται από τον προπολογισμό της ΚΕΠΑ. Θέλουμε όμως επίσης να επαναλάβουμε ένα θετικό στο παρελθόν παράδειγμα, το να δημιουργηθεί ένα, ένα κέντρο ε, για την ε, σχεδίαση, το οποίο θα μπορέσει να συνενώσει χορηγούς από διάφορα κράτη-μέλη που υποστηρίζουν το Μαλί <clears throat> μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας τους. Αυτές λοιπόν οι δυνάμεις, αυτές οι χώρες που δεν θα έχουν ενδεχομένως δυνάμεις ε, στην αποστολή αυτή, αλλά μπορούν να συμμετάσχουν και τρίτα κράτη, με τον τρόπο αυτό δηλαδή μπορεί να υπάρχει χρηματοδότηση, στο παρελθόν χαρη υπήρξε χρηματοδότηση από τον Καναδά για τη χρηματοδότηση παραγωγικά λογισμικού για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων σε μια αποστολή αυτού του είδους. Μπορούμε λοιπόν με τον τρόπο αυτό να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει το κεντρικό, ο κεντρικός αυτός πυρήνας σχεδίασης που θα επιτρέψει να λειτουργήσουν πιο καλά οι επιχειρησιακές μορφές σχεδίασης. Μας δίνει και μεγαλύτερη ευκαμψία για τη δυνητική συμμετοχή τρίτων χωρών. Υπάρχει βέβαια η επίσημη παρουσία <clears throat> εκπροσώπων από τρίτων χωρών. Αυτό δεν ε, είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει για όλα τα κράτη τα τρίτα που ενδιαφέρονται βέβαια, αλλά υπάρχει πάντα η δυνατότητα να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση. Αυτή είναι μια ιδέα που έχουμε αναπτύξει, η οποία μπορεί να δώσει και νέα όθηση στην πολιτική μας για την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων στα πλαίσια αυτών των πολιτικών αποστολών. Τελευταίο σημείο σε ό,τι αφορά τους πόρους. Ενδεχομένω ενδεχομένως ενδιαφέρεται η Επιτροπή σας να γνωρίζει ότι έχουμε εργαστεί σε στενή συνεργασία με την ε, Ευρωπαϊκή Δύναμη Χωροφυλακής. Υπήρξαν εμπειρογνώμονες αυτής της δύναμης που έχουν ε, διαβουλευτεί με τους δικούς μας ειδικού για την ανάπτυξη αυτής της αποστολής και έχει αποφασίσει αυτή η Ευρωπαϊκή Δύναμη Χωροφυλακής να συμμετέχει σε αυτή την αποστολή και θα έχουμε λοιπόν εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα αναπτυχθούν για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν την σωστή κατάρτιση της ε, εθνοφρουράς και της ε, χωροφυλακής στο Μαλί. Και αυτό είναι ένα νέο στάδιο λοιπόν για την ανάπτυξη των σχέσεών μας με την Ευρωπαϊκή Δύναμη <clears throat> Χωροφυλακής. Αναφερθήκατε επίση, κύριε Πρόεδρε στο θέμα της περιφερειακής διάστασης αυτής της αποστολής είναι ένα ερώτημα το οποίο μπορούμε να θέσουμε στον εαυτό μας, κατά πόσο μπορεί να μια περιφερειακή στρατηγική να υλοποιείται μόνο με εθνικές αποστολές. Μια πρώτη απάντηση είναι ότι αυτή τη στιγμή οι παράμετροι και οι περιορισμοί για κάθε χώρα της περιοχής είναι διαφορετικές. Αυτό είναι μια δυσκολία που αντιμετωπίσαμε όταν ξεκινήσαμε την πολιτική αποστολή στον Ήγηρα. Το επίπεδο προόδου το επίπεδο πολιτικής συνειδητοποίησης για την ανάγκη μεταρρύθμισης των δυνάμεων ασφαλείας δεν είναι το ίδιο όταν πρόκειται για τον Ήγηρα, τη Μαυριτανία, το Μαλί κτλ. Υπάρχει λοιπόν ένα κοινό πρόβλημα, αλλά αυτό δεν μπορεί να λυθεί με την <clears throat> ίδια πάντα λύση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την ευκαμψία για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα αυτές τις καταστάσεις που αντιμετωπίσουμε. Μια δεύτερη εξήγηση Υπάρχει και μια πολιτική παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Το γεγονός ότι οι συνομιλητές μας σε αυτή την περιοχή μας το έχουν εξηγήσει ότι θα αντιμετώπιζαν δυσκολίες να έχουν στο έδαφος τους μια αποστολή που θα έχει το δικητήριό της σε μια γειτονική χώρα οι αρχές του Μαλή θέλουν να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχει πλήρης εμπλοκή και έλεγχος από τη δική τους πλευρά και γι' αυτό το λόγο θέλουν αυτή η αποστολή που θα ενισχύσει την εσωτερική ασφάλεια του Μαλή να εδράζεται στο Μαλή και όχι στον Ιγύρα. Αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο το οποίο χρειάζεται να λάβουμε υπόψη. Δεν σημαίνει ότι αυτή η περιφερειακή διάσταση είναι κάτι το οποίο το λησμονούμε. Υπάρχει με δύο πτυχές σε στρατηγικό επίπεδο γιατί οι δράσεις μας εγγράφονται σε μια συνολική στρατηγική για τις χώρες του Σαχέλ και δεύτερον αυτή η περιφερειακή διάσταση υπάρχει λόγω των μηχανισμών συντονισμού και συνεργασίας που έχουμε θεσπίσει μεταξύ όλων των αποστολών στο Σαχέλ και επίσης των αποστολών στο Σαχέλ και της αποστολής στη Λιβύη. Και έτσι η αποστολή ΕΟΚΑΠ στον Ήγηρα έχει διευκολύνει την επαφή το, της αποστολής μας στη Λιβύη με τις αρχές του Νίγηρα για να αντιμετωπιστεί η συνοριακή προβληματική μεταξύ των χωρών αυτών. Τον έχουμε λοιπόν χωριστές αποστολές δεν σημαίνει ότι έχουμε απομονωμένες αποστολές. Προφανώς όμως ζητά μια αυξημένη προσπάθεια συντονισμού και αυτό το έχουμε στο μυαλό μας και φυσικά και η αποστολή πολιτική στο Μαλί. Αυτά λοιπόν θέλω να σας πω για την πρόοδο αυτού του εγχειρήματο και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν παρεμβάσεις. Ε, κυρία Λέζινγκ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λενουάρ. Το γεγονός ότι μιλάμε για το Μαλί δείχνει ότι τα προβλήματα αυτής της περιοχής παραμένουν. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις, πληροφορίε πληροφορίες που μας δώσατε και έχω πολλά ερωτήματα. Είπατε ότι ο στόχος είναι βελτίωση του κράτους δικαίου, της εσωτερικής ασφάλειας, της λειτουργίας του, των εσωτερικών δυνάμεων ασφαλείας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. Και η αποστολή για την οποία αναφέρατε συνεργάζεται με τη Μινούσμα, την αποστολή του ΟΗΕ. Το ερώτημα μου τώρα είναι το εξή. Ποια είναι η εκτίμησή σας για το κατά πόσο όλοι αυτοί οι στόχοι, το κάτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. μπορούν να επιτευχθούν. Εγώ έχω διαβάσει κάποιες εκθέσεις από εκπροσώπους, από μέλη της Μινούσμα, ότι αντιμετωπίζουν εξεγέρσεις στο βόρειο τμήμα του Μάλι. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό και θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η δική σας εκτίμηση για την κατάσταση εκεί και κάποια ερωτήματα για την κατάσταση στο Μαλί. Είναι πολύ δύσκολο για κάποιον απ' έξω να αξιολογήσει αυτή την κατάσταση. Πώς είναι λοιπόν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Τι γίνεται με τις συνομιλίες ειρήνευσης μεταξύ της κυβέρνησης και των ανταρτών. Τι γίνεται στην πόλη Χιντάλ, παραδείγματος χάρη εξακολουθεί να είναι υπό τον έλεγχο των ανταρτών. Και πώς προχωρεί ο αφοπλισμός των ανταρτών. Και αυτό είναι κάτι που έχει μεγάλη σημασία για την επιτυχία της αποστολής. Έχω ακούσει ότι όπως και στο Αφγανιστάν υπάρχει το πρόβλημα της ε, κατά κάποιο τρόπο λιποταξίας στρατιωτών οι οποίοι από τη στιγμή που εκπαιδεύονται φεύγουν και πηγαίνουν σε άλλες ομάδες οι οποίες πρόσκυνται στους αντάρτες. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Και επίσης για την ομάδα αυτή σχεδίου, το, το, την κεντρική μονάδα για τη σχεδίαση αυτό είναι σε εμβριακό στάδιο ή όχι και θα θέλαμε ίσως ενδεχομένως να ξέρουμε ποιες είναι οι τρίτες χώρες οι οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να συνεργαστούν και κατά πόσο μπορούν να δώσουν μια απτή βοήθεια με αυτό το μηχανισμό συντονισμού. Merci. Σας ευχαριστώ. Ζέμκι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Λενουάρ για την ε, ενημέρωση. Και έχω και πολλά ερωτήματα. Πρώτο. Είπατε ότι είστε στην φάση της συγκέντρωσης ε, του ανθρώπινου δυναμικού. Γύρω στα 500 ε, άτομα θα στελεχώσουν αυτή την πολιτική αποστολή. Πώς θα τους επιλέξετε τους εμπειρογνώμονες από πού θα προέρχονται. Θα είναι από το εθνικό επίπεδο, από τα κράτη-μέλη θα προέρχονται και από ποια πλην της Γαλλίας. Δεύτερον, έχετε ένα χρονοδιάγραμμα για αυτήν την αποστολή. διότι πρόκειται και για αρκετά μεγάλο προπολογισμό. Τρίτο ερώτημα. Σχετίζεται και με το ερώτημα της προλαλή σα συναδέλφου. Εκτό των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συμμετάσχουν και άλλε χώρε από την Αφρική. Κυρίω. Ευχαριστώ, Τσάρλ Στάνοκ. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ το έργο της αποστολής στο Μαλί, ήμουν του Κοινοβουλίου για το Σαχέλ και είχα να πω καλά λόγια. Προφανώς πρόκειται για ένα απαραίτητο μέτρο έπρεπε να ληφθεί και φαίνεται ότι πέτυχε και τους άμεσους στόχους ό,τι αφορά την ασφάλεια και τη σταθερότητα στο βόρειο τμήμα της χώρας. Μιας χώρας που είναι ε, που αντιμετωπίζει έντονο κίνδυνο από τους ε, τζιχαντιστές και μπορεί να μεταδοθεί και σε άλλες χώρες ή ε, από τη Σομαλία να υπάρξουν προβλήματα. Συμφωνώ με αυτό που είπε ο Πολωνός συνάδελφος και θέλω και εγώ να επεκταθώ σε αυτό. Πιο ευρωσκεπτικιστές συνάδελφοι μιλάνε για αυτή την αποστολή, λένε ότι οργανώνεται κυρίως από τη Γαλλία και ίσως και βολεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτόν τον τρόπο λόγω έλλειψη σπόρων. Ποια είναι λοιπόν τα άλλα κράτη που θα συμμετάσχουν σε την αποστολή με δυνάμεις, με προσωπικό υπηρογνώμης. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και κάποιοι γλωσσικοί περιορισμοί γιατί ανήκει στη γαλλόφωνη κοινότητα το Μαλί και σίγουρα χρειάζεται η γνώση της γαλλικής γλώσσας. Είναι ένα από τα προσόντα για τα μέλη της αποστολής, ιδίω για μια εκπαιδευτική αποστολή, γιατί δεν είναι εύκολο να έχει κανείς τις υπηρεσίες ενός διερμηνέα. Ποια άλλα κράτη-μέλη συμμετέχουν και αν υπάρχει, ποια είναι η συνεργασία, ο συντονισμός και η διασύνδεση με την Αφρικανική Ένωση και το ΕΚΟΒΑΣ. Θα υπήρχε ανάπτυξη μιας ε, αποστολής από το ΕΚΟΒΑΣ. Φαντάζομαι, επειδή μιλήσατε για την ψήφιση των Ηνωμένων Εθνών, έχετε επαφή με τον ΟΗΕ για την ε, θέσπιση της νομικής βάσης. Αλλά με τις δομές της Αφρικανικής Ένωσης, της Αφρικανικής Πύρων Γέννη, τι συνεργασία υπάρχει, Πρόεδρος. Άλλες παρεμβάσεις, όχι, κύριε Γενική Διευθυντά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλες αυτές τις ερωτήσεις. Θα έπρεπε ίσως ορισμένα από αυτά με ρωτάτε τα, να τα είχα αναφέρει στην εισαγωγή. Και ιδίως αυτό το ζήτημα της, του συντονισμού με τον ΟΗΕ. Έχουμε εργαστεί πάνω σε αυτό το θέμα και επί το, με τον κύριο Κούντερς στη Νέα Υόρκη, με τους ε, συνομιλητές μας από το DPTO. Τι κάνουμε λοιπόν. Ουσιαστικά θέλουμε να συμπληρώσουμε το έργο των Ηνωμένων Εθνών. Δεν θέλω να ψέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά σχηματικά αποφασίσαμε τα Ηνωμένα Έθνη λόγω της δικής τους εντολής διατηρούν τη γενική ευθύνη και αρμοδιότητα για τη μεταρρύθμιση των εθνικών δυνάμεων ασφαλείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάσσεται στο πλαίσιο αυτό και αναλαμβάνει κάποια συγκεκριμένα καθήκοντα. Τα Ηνωμένα Έθνη επίσης θα έχουν υπό την ευθύνη τους την πιο άμεση υποστήριξη στη δικαιοσύνη. Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, προσπαθούμε να διαρθρώσουμε τη δική μας δράση. Ξέρετε ότι δεν είναι οι ίδιοι μηχανισμοί λήψη αποφάσεων, ούτε είναι και οι δομέ ίδιε. άρα αυτή η εργασία συντονισμού απέτησε μεγάλη προσπάθεια. Πιστεύω όμω ότι τώρα έχουμε ένα μηχανισμό που κατά την άποψή μου είναι καλά διαρθρωμένος ε, σε σχέση με τον ΟΗΕ. Ο άλλος μας εταίρος που αναφέρατε και εσείς είναι η Αφρικανική Ένωση. Η Αφρικανική Ένωση είναι παρούσα, έχει πολιτική παρουσία επιτόπου ε, και διαχείριση ε, κρίσεων που ήταν δική της αρμοδιότητα, πλέον αρμοδιότητα των Ηνωμένων Εθνών. Εμείς παρουσιάσαμε τις ιδέες μας στην Αφρικανική Ένωση ώστε να είναι ενήμεροι για το τι εμείς κάνουμε, αλλά το ζήτημα του συντονισμού με την Αφρικανική Ένωση από τη στιγμή που δεν έχει κάποια συγκεκριμένη δέσμευση δεν τίθεται με τους ίδιους όρους, όπως δηλαδή με τα Ηνωμένα Έθνη. Η κυρία Λέζη μίλησε, με, μίλησε για τη σχέση με ε, τις πολιτικές διαδικασίες. Δεν είμαι σχετικά ειδικό, άρα δεν μπορώ να απαντήσω διεξοδικά, αλλά νομίζω ότι αυτό που ουσιαστικά υπονοούσατε είναι αν αυτά που εμείς κάνουμε έχει νόημα αν δεν υπάρχει πολιτική διαδικασία. Η απάντηση που μπορώ να δώσω στην ερώτησή σας είναι φυσικά ότι αυτό που οι δικές μας αποστολές είναι σε θέση να κάνουν στο δικό τους επίπεδο μπορούν να πετύχουν, να έχουν συγκεκριμένα αυτά αποτελέσματα παρά μόνο αν υπάρχει μια πολιτική διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης που θα φέρει και καρπούς. Αυτή είναι η λογική και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έχουμε αυτή τη στρατηγική για το Σαχέλ. Έχουμε την πολιτική ε, συμφιλίωση, ε, την εθνική συμφιλίωση και πιο συγκεκριμένες όμως δεσμεύσεις ε, για τις δυνατότητες στρατιωτικές και μη. Μιλήσατε για ένα δύσκολο, δύσκολο ζήτημα τα prerequisites, τα προαπαιτούμενα όπως τα λέμε, δηλαδή αυτοί που εκπαιδεύουμε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε τις δυνατότητες και ικανότητες που θα αποκτήσουν δεν θα τις χρησιμοποιήσουν εναντίον μας. Πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό στην περίπτωση της εκπαίδευσης και δημιουργίας υποδομών. Το ε, θέμα μας απασχόλησε στην Σομαλία. Δηλαδή θέλαμε οι στρατιώτες που εκπαιδεύουμε να παραμείνουν στις δικές μας μονάδες και να παραμείνουν υπό τον έλεγχο των νόμιων πολιτικών αρχών. Γι' αυτό το λόγο αυτή η εκπαιδευτική δράση δεν θέλαμε να είναι απομονωμένη. Θελήσαμε αντίθετα αυτή η εκπαιδευτική αποστολή να συνοδεύεται από εργασία στο πλαίσιο της αλυσίδας διοίκησης που θα λειτουργεί. Και αυτοί ε, οι άνθρωποι να τεθούν υπό την αιγίδα αυτής της ε, διοίκησης και να υπάρχει λογοδοσία στις πολιτικές δικαστικές αρχές, του Μαλή συγκεκριμένα. Δεν μπορώ να σας εγγυηθώ 100% ότι όλοι οι αστυνομικοί του Μαλή θα παραμείνουν στις μονάδες τα κτλ. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε πλήρη αλυσίδα που επιφέρει τις στις δυνατές εγγύσεις να είναι επιτόπου. Και αυτή είναι η εντολή που έχουμε. Είμαστε στη φάση της διαχείρισης κρίσης, δεν μπορώ να σας δώσω δυστυχώς εγγύσεις 100% ότι έτσι θα ε, εξελιχθούν τα πράγματα. Αλλά μπορώ να σας εγγυηθώ ότι θα κάνουμε πάντο δυνατόν και το έχουμε ήδη κάνει για να πετύχει αυτή η αποστολή. Μιλήσατε για τις τρίτες χώρες, ως ήθιστές, τις αποστολές ΕΠΑ, Πολλές τρίτες χώρες ε, μπορούν να συμμετέχουν, δεν έχω τον κατάλογο. 20 και πάνω χώρες ε, έχουν κληθεί να συμμετάσχουν. Έχουμε τους συνήθεις εταίρους φυσικά, τις ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Αμερικανοί, Καναδοί, φίλοι, Νορβηγοί φίλοι, επίσης οι χώρες με τις οποίες ήδη έχουμε συνεργασία στα θέματα άμυνας και ασφάλειας, χώρες με τις οποίες έχουμε συνάψει συμφωνίες συμμετοχής. Αλλά θα μπορούσα μέσω της γραμματείας της Επιτροπής σας να σας διαβιβάσω τον ακριβή κατάλογο των χωρών. Αλλά υπάρχει αυτή η ανάγκη να έχουν συμμετοχή και τρίτες χώρες και την έχουμε λάβει υπόψη μας. Θέσατε επίσης το ερώτημα ε, πραγματικής ευρωπαϊκής αποστολής, έτσι εγώ το καταλαβαίνω το ερώτημα, απέναντι ε, στο να είναι αυτή η αποστολή, έναντι μάλλον του να είναι αυτή η αποστολή καθαρά γαλλική. Αρκεί να δείτε αυτή την παιδευτική αποστολή στο Μαλί για να καταλάβετε ότι ναι μεν αυτή την ιδέα την πρόθεσαν οι Γάλλοι αρχικά, αν και πάλι δεν συμφωνώ ότι έτσι είχαν τα πράγματα, ήταν τέτοια κατάσταση ασφάλεια στο Σαχέλ, ιδίω μετά τα γεγονότα της περσινής χρονιάς, ομοιρία στην Αλγερία. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν πραγματικά ε, ενδιαφέρον και συμφέρον να είναι ασφαλής η περιοχή του Σαχέλ και πέραν τη αναπτυξιακή βοήθεια και τη πολιτική δέσμευση, πολλοί θεωρούν ότι θα πρέπει να συμπληρώσει αυτή τη δέσμευσή τη η Ευρωπαϊκή Ένωση με δέσμευση και στον τομέα τη άμυνα και ασφάλεια. Την πολιτική αποστολή στο Μάλι δεν νομίζω ότι μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε ως μια αποστολή που προώθησε, θέλησε και τελικά στελεχώνει μόνο η Γαλλία. Δεν μπορώ σήμερα να σας δώσω τον κατάλογο των χωρών που θα συμμετέχουν γιατί δεν έχουμε ακόμη αρχίσει ε, να οργανώνουμε και να συνθέτουμε αυτή την αποστολή. Θα είναι και άλλες όμως χώρες που θα συμμετέχουν. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όταν δει κανείς την εκπαιδευτική αποστολή στο Μαλή βλέπει και έτσι βλέπουμε ότι και η σκητάλη θα, είναι, θα την πάρει μια πολυεθνική αποστολή. η ευρωπαϊκή δέσμευση στο Μαλή νομίζω ότι είναι πολύ πιο πολύ γενική παρά εθνική που πήρε μετά και έτσι τα ευρωπαϊκά χρώματα. Ένα άλλο στοιχείο που θα έπρεπε να είχα αναφέρει όταν ε, έκανα την εισαγωγή μου είναι το χρονοδιάγραμμα. Δική μας εκτίμηση είναι ότι για να πετύχουμε τους στόχους που ορίσαμε για αυτήν την αποστολή και τους οποίους δέχονται και τα κράτη-μέλη, απαιτούνται τέσσερα χρόνια. Στόχος μας είναι να έχουμε μια αρχική εντολή δύο ε, χρόνια και μετά ενδιάμεσα δηλαδή να δούμε τι πρόοδο έχουμε επιτελέσει και ιδίω στο κατά πόσον ιδιοποιούνται τη διαδικασία αυτή οι αρχές του Μαλή. Γιατί θα έχει νόημα αυτή η τετραετή προσπάθεια εάν την αναλάβουν, την ιδιοποιηθούν στη συνέχεια οι αρχές του Μαλή. Εκτιμούμε λοιπόν από πλευρά σχεδιασμού προγραμματισμού ότι για να πετύχουμε τα αποτελέσματα τα ευκταία ε, μας χρειάζονται τέσσερα χρόνια. Ζητήσαμε όμως μια αρχική εντολή δύο ετών με ρήτρα αναθεώρησης για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε εάν και κατά πόσον θα επιμικίνουμε ε, για δύο χρόνια ακόμη. Και στο Κονγκό είχαμε αυτό, το, την ομάδα ε, σχεδίων. Ε, δεν είναι κάτι καινούριο, θα το υιοθετήσουμε και στην περίπτωση του Μαλή. Έχει δύο καινούριες πτυχέ. Αυτή η μονάδα έργων, σχεδίων συμπληρώνει ένα κενό προηγούμενων αποστολών σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση εξοπλισμού ασφαλείας οι κανόνες και οι μηχανισμοί που ισχύουν καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή τη χρηματοδότηση εξοπλισμών για τις δυνάμεις ασφαλείας. Με αυτό το νέο, λοιπόν, αυτή τη νέα μονάδα θα μπορούμε να έχουμε αυτή τη χρηματοδότηση για να καλύψουμε αυτά που δεν μπορούμε να καλύψουμε με άλλα μέσα. Και δεύτερος στόχος είναι να παράσχουμε σε τρίτες χώρες τη δυνατότητα εταιρικής σχέσης που δεν θα συνεπάγεται κατά ανάγκη ότι θα πρέπει να συμμετάσχουν ε, πλήρως σε μια ευρωπαϊκή αποστολή. Σε ό,τι αφορά την εκπαιδευτική αποστολή στο Μαλί, ο Καναδάς για παράδειγμα για λόγους ασφαλείας δεν επιθυμούσε ανάπτυξη με στρατεύματα ε, στο Μαλί. Ήθελε όμως, επειδή συμμεριζόταν τις ε, δικές μας ανησυχίες, να έχει μια συμμετοχή Όσοι λοιπόν συμμερίζονται τους στόχους μας αλλά για εθνικούς δικούς τους λόγους δεν θέλουν να αναπτύξουν ε, ε, στρατιωτικές δυνάμεις έχουν αυτή τη δυνατότητα. Δεν είναι λοιπόν κάτι καινούριο. Μπορούμε να ε, έχουμε αρχίσει να το εφαρμόζουμε και από παλιότερα. Ελπίζω να έχω απαντήσει όλα τα ερωτήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις από άλλους συναδέλφους. Δεν βλέπω κανέναν. Θα συνεχίσουμε πάντως να παρακολουθούμε όλες αυτές τις εξελίξεις και σας ευχαριστούμε αν μπορείτε πράγματι να έρχεστε εδώ πέρα και να μας ενημερώνετε για τις περαιτέρω εξελίξεις. Η κυρία Λέζινγκ αναφέρθηκε στο ότι όντως χρειαζόμαστε μία τακτική ενημέρωση όσον αφορά το Μαλί και κατά τη διάρκεια της όλης εντολής της αποστολής εμείς εστιαστήκαμε πάρα πολύ στην περιοχή του Σαχέλ που μέσω τουλάχιστον των κειμένων που έχουν εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα της λεγόμενης σφαιρικής ολιστικής προσέγγισης για μια περιφερειακή στρατηγική. Ακούστηκαν βέβαια κάποιες επικρίσεις για το ότι ήταν ιδιαίτερα βραδία η εφαρμογή και η ανάπτυξη της στρατηγικής αυτής, αλλά βλέπουμε πλέον ότι αρχίσουμε και να αναπτυσσόμαστε με έναν τρόπο πολύ πιο γρήγορο, προκαθορισμένο και σας συγχαίρουμε λοιπόν γι' αυτό Θεωρώ πάντως ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε προκειμένου να καταφέρουμε να εξορθολογήσουμε καλύτερα τα διαθέσιμα μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε. Και είπατε κι εσείς ότι ένα πρόβλημα το οποίο παραμένει είναι να δούμε πώς θα καταφέρουμε στα πλαίσια μιας περιφερειακής στρατηγικής να χρησιμοποιήσουμε εθνικά μέσα. Πώς μπορούμε εμείς από ευρωπαϊκής πλευράς να βελτιστοποιήσουμε τα εθνικά αυτά μέσα, πώς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε την αποστολή αυτή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε όλη την οργανωτική πλευρά της αποστολής. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να επαγρυπνήσουμε για όλα αυτά τα ζητήματα, μολονότι νομίζω ότι επί της αρχής μπορούμε να σας συγχαρούμε για το ότι βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όλο και περισσότερο είναι παρούσα και προσπαθεί να επιλύσει τα προβλήματα της περιοχής αυτής, τα οποία βέβαια ακόμα παραμένουν ανεπίλητα. Βλέπουμε επίσης ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία επηρεάζουν και άλλες περιοχές πλέον στην Αφρική. Πολλές φορές εστιάζουμε τελευταία την προσοχή μας σε άλλες περιοχές ε, της Αφρικής και όχι τόσο πολύ στο Μαλί, ενώ πιστεύω ότι θα πρέπει να μην ξεχνάμε και την περίπτωση του Μαλί, όπου από πολιτικής, διπλωματικής και στρατικής πλευρά έχουμε μια σημαντική παρουσία. Να περιμένουμε λίγο και τη συνάδελφο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως θα μας μιλήσει για ζητήματα ασφάλειας στην θάλασσα. Την ε, επόμενη εβδομάδα θα υπάρχουν επαφές με εκπροσώπους της Αφρικανικής Ένωσης ε, από πλευράς ε, κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Πιστεύετε ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να θίξουμε. Μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα σε σχέση με τις επαφές που έχετε με τους αδέλφους από την Αφρικανική Ένωση, ιδίως όσον αφορά τον εντεταλμένο για ζητήματα ειρήνης απάντηση. Κοιτάξτε, έρχεται την κατάλληλη στιγμή η ερώτηση αυτή, γιατί όντως πλησιάζει σύνοδος της Αφρικανικής Ένωσης και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της εβδομάδος αυτής θα αναφερθεί και στο ζήτημα των σχέσεων που έχουμε με την Αφρικανική Ένωση, ιδίως το ζήτημα της συνεργασίας μας σε ζητήματα ασφάλειας. Ποια είναι η δική μας τώρα η άποψη, η δική μας η προσέγγιση. Υπάρχει μια έντονη άμεση αλληλοσυμπληρωματικότητα. Η βασική ιδέα είναι να καταφέρουμε να διασφαλίσουμε αφρικανικές λύσεις στα αφρικανικά προβλήματα. Εμείς είμαστε απλώς εταίροι που θα βοηθήσουμε τους Αφρικανούς να εφαρμόσουν τις λύσεις αυτές η διαμόρφωση της όλης αρχιτεκτονικής ειρήνευσης ε, και ασφάλειας στην Αφρική είναι κάτι το οποίο αποτελεί και δική μας πρόθεση και δικό μας στόχο. Δεύτερον, η Αφρικανική Ένωση όσον αφορά τη διαχείριση των κρίσεων. Κατάφερε να δείξει ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Η ΣΟΜ, για παράδειγμα, αποτελεί, νομίζω, την καλύτερη προστιθέμενη αξία των αφρικανικών μέσων τα οποία χρησιμοποιούνται για την εγκαθίδρυση της ε, ειρήνης. Νομίζω ότι αν δεν είχαμε την αμισόμα δεν θα καταφέρναμε να είχαμε την κατάσταση που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Σομαλία και αν δεν είχαμε τη συμβολή των, ε, και τη θυσία που, έκανε οι Αφρικανικές χώρες δεν θα είχαμε τα θετικά αυτά αποτελέσματα στα πλαίσια της αμισόμ. Θεωρώ πάντως ότι η δική μας η προσέγγιση όσον αφορά την αρχιτεκτονική ε, ειρήνης και ασφάλειας στην Αφρική Υπάρχει μία ευκταία ισορροπία την οποία πρέπει να πετύχουμε. Από τη μια πλευρά πρέπει από θεσμικής πλευράς να υποστηρίζουμε τα θεσμικά όργανα της Αφρικής. Υπάρχει λοιπόν αυτή η θεσμική υποστήριξη προς τις αφρικανικές αρχές από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ επίση και στι διάφορε περιφέρειε και υποπεριφέρειε και θέλουμε επίση να υποστηρίξουμε και τι διάφορε ε, εθνικέ ε, αρχέ ε, ασφάλεια. Καταλαβαίνετε όμως ότι η δική μας η συμβολή δεν έχει κανένα νόημα αν δεν υπάρξει και συμβολή από την αφρικανική πλευρά. Δεν θα έχουμε αποτελεσματική ειρήνευση στην Αφρική αν δεν υπάρχει και η συμβολή των ε, αφρικανικών δυνάμεων. Γι' αυτό και στα πλαίσια αποστολών όπως η UTM ή στα πλαίσια των αποστολών που μόλις τώρα καλύψαμε, στόχος μας είναι να καταφέρουμε να αλλοσυμπληρώσουμε, να συμπληρώσουμε μάλλον εμείς, τις προσπάθειες που ήδη γίνονται από τις εθνικές αφρικανικές αρχές ασφαλείας. Αυτή άλλωστε την εντολή μας έχει δώσει και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που μετά από γερμανική πρόταση μας ζητήθηκε να καταφέρουμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας και τη δέσμευσή μας σε σχέση με τα εθνικά συστήματα ασφάλειας των Αφρικανικών κρατών. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι ένα από τα βασικά ζητήματα που θα μας απασχολήσει στο μέλλον με την Αφρικανική Ένωση να καταφέρουμε να βρούμε την καλύτερη αυτή δυνατή διάρθρωση. Δηλαδή, πώς θα καταφέρουμε να συνδυάσουμε τη δική μας συμβολή με τη συμβολή των Αφρικανικών αρχών και πώς μπορούμε εμείς να βελτιώσουμε μέσω της δικής μας συμβολής τα αποτελέσματα του έργου των Αφρικανικών δυνάμεων. Ήδη χρησιμοποιούμε κάποια μέσα, κάποια εργαλεία. Έχουμε τις αποστολές ΚΕΠΑ, καθώς επίσης και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας. Θα μπορούσαν όμως τα μέσα αυτά να συμπληρωθούν και με άλλα εργαλεία και με άλλα μέσα, προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε μια σφαιρική προσέγγιση τη της ανάπτυξης των εθνικών αυτών μέσων. Νομίζω ότι κάτι το οποίο πρέπει να αποφύγουμε είναι να θεωρήσουμε ότι η ανάπτυξη των εθνικών αυτομέσων έχει να κάνει μόνο με την εκπαίδευση και την κατάρτιση δεν αρκεί να καταρτήσουμε απλώς κάποιες στρατιωτικές μονάδες, δεν έχουμε βελτιώσει την, το, το γενικότερο καθεστώς των εθνικών αυτών αρχών. Έχουμε βελτιώσει κατά κάποιο τρόπο μόνο την αποτελεσματικότητα των δυνάμεων αυτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να δούμε και όλες τις υπόλοιπες πλευρές και τις μη στρατιωτικές πλευρές. Το νομικό πλαίσιο, το αστυνομικό πλαίσιο, το γενικότερο εθνικό πλαίσιο το οποίο ισχύει στις χώρες αυτές. Είναι Πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το πετύχουμε αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό το έχουμε αυτό κατά νου κάθε φορά που μιλάμε για σφαιρική ολιστική προσέγγιση όσον αφορά τη συνεργασία μας με τις Αφρικανικές Αρχές. Πρόεδρος, και για να ολοκληρώσουμε για το ζήτημα αυτό, όσον αφορά την γεωγραφική διάσταση, νομίζω που πρέπει ακριβώς να δώσουμε βάρος στη Σομαλία, στο Μαλί, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Κοιτάξτε, όντως αναφέρθηκα σήμερα σε διάφορους τομείς συνεργασίας. Προφανώς υπάρχει συνεργασία στην Σομαλία, όπου υπάρχει όλο και καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στις διάφορες αποστολές μας. Βασιζόμαστε στις πολύ, στα πολύ καλά αποτελέσματα που είχαμε στα πλαίσια της Αμισόμ και ακριβώς αυτά προσπαθούμε να εφαρμόσουμε και στα πλαίσια της e UTM. Εμείς εκπαιδεύουμε ουσιαστικά τους στρατιώτες, αλλά είναι η Αμισόμ στη συνέχεια που χρησιμοποιεί τους στρατιώτες αυτούς στην Μογκαντισού προκειμένου να τους χρησιμοποιήσει επιτόπου. Αυτό λοιπόν κάναμε στη Σομαλία. Έχουμε μια πιο, όλο και πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. Στην αποστολή μας αυτή μας βοηθάει και η Αφρικανική Ένωση στα πλαίσια της Αμισόμα. Στο Μαλί αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα πέρα από την εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι η γενικότερη αναδιοργάνωση των δυνατοτήτων άμυνας στο μέλλον, όχι τώρα, αλλά κάποια στιγμή στο μέλλον, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να επιφέρουμε κάποιες γενικότερες μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση άμυνας που υπάρχει στη Σομαλία, πώς μπορούμε να εμπλέξουμε και περισσότερες μονάδες. Εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε πάντως την Αφρικανική Ένωση να αυξήσει τις δυνάμεις της και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια στον Μπαγκή με την Αφρικανική Ένωση. Η κυρία Ζουμά ε, πρόσφατα ε, έστειλε μια επιστολή στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, λέγοντας ότι υποστήριζε την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής αποστολής στη χώρα. Θεωρώ λοιπόν θα μπορούσαμε και στα πλαίσια της συνεργασία αυτής να είχαμε θετικά αποτελέσματα. Όσον αφορά τώρα το Μαλί και τη γενικότερη περιοχή του Σαχέλ, Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας πολιτικός διάλογος. Η Αφρικανική Ένωση μέχρι στιγμής δεν έχει συγκεκριμένη αποστολή ε, διατήρηση της ειρήνης ε, στην χώρα αυτή. Διεξάγεται ένας διάλογος ο οποίος είναι περισσότερο πολιτικός και όχι τόσο επιχειρησιακός. Στο μέλλον πάντως ε, θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορούσε και στην περίπτωση αυτή η Αφρικανική Ένωση να συμμετάσχει περισσότερο. Βέβαια υπάρχουν περιορισμοί όπως το ξέρετε ε, ότι πρέπει κάθε φορά με βάση τη γεωγραφική περιοχή στην οποία αναπτυσσόμαστε να λάβουμε υπόψη μας και τις ε, περιφερειακές ιδιαιτερότητες. Πάντως εξετάζουμε και αυτή την εναλλακτική λύση, Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτές τις διευκρινήσεις σε σχέση με τις αφρικανικές δυνάμεις. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημέρας τη διάταξης, που είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας για την ασφάλεια στη θάλασσα. Είπαμε προηγουμένω ότι είναι μία από τις πιο φιλόδοξες προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου για τα θέματα ασφάλειας και άμυνας. Υπάρχει μια ευρύτατη συνένεση μεταξύ των 100 μελών για τα θέματα αυτά, ακόμα και αν βέβαια δεν ε, έχουν την ίδια, α, τις ίδιες προτεραιότητες οι χώρες οι οποίες έχουν ε, μεγάλες ε, ακτογραμμές στην ε, Ευρώπη που έχουν τις ίδιες προτεραιότητες. Πολλές φορές οι προτεραιότητες εστιάζονται στην καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης κτλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντως είναι απαραίτητο να μπορέσει το ταχύτερο δυνατό να έχει μια στρατηγική για την ασφάλεια στη θάλασσα και κυρίως να μπορέσει να εφαρμόσει μια τέτοια στρατηγική. Μπαίνουμε λοιπόν σε ένα ενάρετο κύκλο σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά. Στην επιτροπή μας η κυρία Γκόμες ήταν αυτή η οποία είχε συντάξει μια έκθεση για τα θέματα αυτά που ήταν ιδιαίτερα πλήρης. Φυσικά η ασφάλεια στη θάλασσα περιέχει πάρα πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και ο στόχος μας είναι μαζί και με την κυρία Γκμίντερ να μπορέσουμε, η οποία είναι προστάμενη μονάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με εσάς κύριε Λενουάρ για το θέμα της ΕΠΑ, να μπορέσουμε να κάνουμε μια επισκόπηση της κατάστασης, να δούμε πού βρισκόμαστε, γιατί περνάει ο χρόνος <clears throat> και θα πρέπει να γνωρίζουμε και πού βρίσκονται τα πράγματα πριν από το τέλος της θητείας μας σε σχέση με το έργο που έχει γίνει και με τα χρονικά ορόσημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Θα δώσω καταρχήν το λόγο στην κυρία Γκμίντερ ώστε να μπορέσει να ξεκουραστεί λιγάκι ο κύριος, ε, ο κύριος ε, Λενουά. Μπορώ να μιλήσω γερμανικά. Θα μπορούσα να μιλήσω γερμανικά μάλλον, αλλά δεν ξέρω την ορολογία, γι' αυτό θα μιλήσω στα αγγλικά. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι εδώ ενώπιον σας οι περισσότεροι από εσά θα έχετε ήδη δει ποια είναι τα κύρια στοιχεία της ε, προτινόμενης στρατηγικής για τη θαλάσσια πολιτική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σα τα έχει παρουσιάσει και η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο. Υπήρξε πολύ καλή συνεργασία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και τη Κομισιόν για τη στρατηγική αυτή που δεν είναι ακόμα πλήρω αρθρωμένη γιατί δεν είναι ακόμα σαφή τα στοιχεία τα οποία θα την απαρτίζουν και τα κρατη δεν έχουν δώσει ακόμα σχόλια σε σχέση με αυτή τη στρατηγική. Φυσικά περιμένουμε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμβάλλει και αυτό με τα σχόλιά του. Είναι σαφές από πού ερχόμαστε. Υπήρχε καταρχήν ε, η, τα καθήκοντα τα οποία διατυπώθηκαν επί Ισπανικής Προεδρίας, μετά ακολούθησαν τα σχόλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πολλών κρατών μελών, όπως είναι η Κύπρος, η Γαλλία, η Ιρλανδία, που διατύπωσαν στοιχεία στρατηγικής που ξεφεύγουν μονάχα από την ε, περιοχή της ΕΠΑ και επομένως περιλαμβάνουν και εξωτερικές και εσωτερικές πολιτικές και η έκθεση Γκόμες <clears throat> είναι κάπως στο παρελθόν αλλά πήραμε πολλά σημαντικά μηνύματα από αυτή την έκθεση για να μπορέσουμε να μπορέσουμε συγγνώμη, να καταλήξουμε σε εγκάσιους στόχους και εγκάσια συνεργασία εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών. Η ελληνική Προεδρία έκανε μία από τις εμβληματικές της πρωτοβουλίες την ε, θαλάσσια στρατηγική ασφάλειας και ελπίζουμε ότι στις 20 Ιουνίου θα εγκριθεί αυτή η στρατηγική. Είναι αρκετά φιλόδοξο αυτό το χρονοδιάγραμμα, αλλά δεν είναι και το τέλος της, της διαδικασίας, γιατί η στρατηγική αυτή θα πρέπει να θεσπίσει βασικούς τομείς προβληματισμού, αλλά δεν πρόκειται να έχει δυνατότητα να καθορίσει την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής, θα πρέπει στη συνέχεια να συμφωνήσουμε για τις ενδεχόμενε δράσεις οι οποίες θα πρέπει να αναλυθούν και την εφαρμογή τους. Οι δυνατότητες λοιπόν αυτών των δράσεων είναι πράγματι σημαντικές και ευρείες. Θέλουμε λοιπόν και τις δικές σας κατευθυντήρες γραμμές και τις κατευθυντήρες γραμμές των κατών μελών για να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρα σε αυτό το εγχείρημα, αλλά είναι σίγουρα ένας χώρος εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άμεσο μέλλον και ένα χώρος στρατηγικής σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα βασικά στοιχεία αναφερόμαστε στις απαραίτητες αρχές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ότι πρέπει να αναπτύξουν τις απαραίτητες και κατάλληλες πολιτικές και έχουμε και κάτι το οποίο αναφέρεται για πρώτη φορά, δεν είναι προφανές, για πρώτη φορά αναφέραμε ποια είναι τα ευρωπαϊκά συμφέροντα στο χώρο της θάλασσας αλλά και ποιες είναι και οι απειλές που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο θαλάσσιο χώρο. Μιλάμε για την πρόληψη συγκρούσεων, διατήρηση ειρήνης, ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας με συνεργασία και με διεθνούς, διεθνείς εταίρους. Αναφερόμαστε για την προστασία των κρίσιμων θαλάσσιων υποδομών μας. Ξέρουμε όλοι ότι αυτός είναι σημαντικός στόχος. Αυτό περιλαμβάνει τα λιμάνια, τις ε, υπεράκτιες εγκαταστάσεις, τηλεκοινωνιακά καλώδια κτλ. Υπάρχουν όλα αυτά τα οποία χρειάζονται την προστασία μας. Ουσιαστικό ουσιαστικός, ε, ουσιαστική προστασία των εξωτερικών συνόρων, διατήρηση των ε, αλυσίδων εφοδιασμού και επάταξη της άναρχης και παράνομης αλίας. Όλα αυτά λοιπόν είναι σημαντικά στοιχεία συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε και τις απειλές που είναι εδαφικές διαμάχες για τα χωρικά ύδατα ή τις αποκλειστικές ζώνες. Η ύπαρξη όπλων μαζικής καταστροφής, ε, η πειρατεία, η τρομοκρατία και άλλες παράνομες πράξεις εναντίον ε, επιβατηγών ή φορτηγών πλοίων, το οργανωμένο έγκλημα, η θαλάσσια λαθρεμπορία ναρκωτικών ή όπλων και φυσικά οι δυνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, η απόρριψη ρήπων στη θάλασσα, αποτελέσματα ακραίων ε, γεγονότων και θαλασσίων καταστροφών. Όλα αυτά λοιπόν, τα συμφέροντα από τη μια μεριά και οι απειλέ από την άλλη μεριά, όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν για να δούμε ποιο θα είναι το περιεχόμενο τη στρατηγική μα. Ο στόχο μα είναι να χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τι δυνατότητε οι οποίε υπάρχουν σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό βέβαια επίπεδο και πολλά από τα θέματα τα οποία συζητούμε αυτή τη στιγμή είναι στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Επομένω, αυτή η στρατηγική θα πρέπει να εμπλέξει και τα κράτη-μέλη και να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να δουν με ποιο τρόπο θέλουν να αντιμετωπίσουν και να συνεργαστούν καλύτερα για τα θέματα αυτά στους διάφορους τομείς οι οποίοι εμπλέκονται στην προστασία από τις ε, απειλές ασφαλείας στη θάλασσα, μιλάμε για θέματα τελωνίων, θαλασσίων μεταφορών, αυτά είναι θέματα πραγματικά χάρη Υπουργών Εσωτερικών Υποστασίας του Πολίτη, υπάρχουν θέματα περιβάλλοντος, υπάρχουν θέματα αλίας για την επιθεώρηση της αλίας. Όλα αυτά λοιπόν εμπλέκονται σε αυτό το στόχο. Θέλουμε επίσης να προωθήσουμε, αλλά ο Διντία θα πει περισσότερο, μια ουσιαστική εταιρική σχέση στο θαλάσσιο χώρο. Θέλουμε επίσης να προχωρήσουμε σε ένα πιο αποτελεσματικό σε σχέση με το κόστος τρόπο συνεργασίας. Συνεργαζόμαστε ήδη, μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα στο μέλλον, μπορούμε να το κάνουμε πιο αποτελεσματικά και πολλές από τις δράσεις που αναλαμβάνουν οι δυνάμεις ασφαλείας με σωστή συνεργασία ή σωστή κίνηση σχεδίαση μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Και έτσι να δώσουμε στους πολίτες μας μια καλύτερη μορφή προστασίας. Τέλος, θέλουμε και αυξημένη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και είναι η πεποίθησή μας ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με εγκάρσιες μορφές συνεργασίας σε συνεργασία στρατιωτικών και πολιτικών αρχών. Θέλουμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε μια λειτουργική ακαιρεότητα, δηλαδή ο καθένας διατηρεί τις αρμοδιότητες του και την αποστολή του. Δεν αλλάζει ο τρόπος που λειτουργεί η αποστολή των οργανισμών, αλλά σε σχέση με το τι κάνουμε, στην πράξη να υπάρχει η σωστή συνεργασία. η πολυμέρεια στο θαλάσσιο τομέα είναι πάρα πολύ σημαντική, δεν πρόκειται να πω περισσότερα εδώ και φυσικά ο σεβασμός για τους κανόνες και τις αρχές του διεθνούς, του διεθνού δικαίου, διεθνούς δικαίου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν μας παρουσιάζει τις αρχές, τους στόχους έχουμε και τις απειλές και αυτά οδηγούν σε πέντε δομικούς λίθους που έχετε στο έγγραφό μου. Δεν πρόκειται να περάσω σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Είναι, η, <clears throat> είναι προς το παρόν προτάσεις, συστάσεις από την πλευρά των κρατών μελών. Πρώτον, εξωτερική συνεργασία. Δεύτερον, ε, διαμοιρασμός πληροφορίας για τα θαλάσσια θέματα. Γιατί μπορούμε να κερδίσουμε πολλά από την ε, θέση σε κοινού των πληροφοριών που έχουμε μπορεί να οδηγήσει σε μείωση κόστους για να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη για τη συλλογή δεδομένων και στη συνέχεια στο επόμενο βήμα μπορεί να υπάρχει κοινό σχεδιασμός δραστηριοτήτων. Ένα καλό παράδειγμα είναι αυτά τα οποία έγιναν πέρσι μετά το, την τραγωδία της Λαμπεδούσα οι χώρες της Μεσογείου, κυρίως η Ιταλία, έφτιαξαν ένα σχέδιο για το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τους πόρους μας στη Μεσόγειο. Όταν υπάρχει ένα πλοίο, παραδείγματος χάρη του ναυτικού ή του, ε, του, τε, των τελωνιακών αρχών, να μπορεί να συνεργάζεται με τους άλλους για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Τρίτο στοιχείο είναι διαχείριση κινδύνου και προστασία κέριων υποδομών και επίσης και <clears throat> έρευνα και ανάπτυξη, καινοτομία και δημιουργία ικανοτήτων, τη εκπαίδευση κτλ. Έχουμε λοιπόν κάθε εμπιστοσύνη ότι με αυτή τη στρατηγική για τα θαλάσσια θέματα, που είναι η πρώτη που αναπτύσσεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τα κράτη-μέλη έχουν στρατηγικές, αλλά είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια συνολική στρατηγική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχει μια κοινή πολιτική, να είναι πιο αποτελεσματική, να έχει καλύτερη εταιρική σχέση και να προστατεύει καλύτερα του πολίτες μας. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Λενό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τελικά δεν έχω και πολλά να προσθέσω στην προηγούμενη παρουσίαση. Να υπενθυμίσω ίσως το γενικό πλαίσιο στο οποίο θέλησαμε να εντάξουμε αυτήν την εργασία μας για την ανάπτυξη της θαλάσσιας στρατηγικής. Θέλαμε να συμπεριλαμβάνει όσο δυνατόν περισσότερα πράγματα αυτό το πλαίσιο. Εσείς αναφέρατε και την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε, και σαφώς αυτό το έγγραφο μας καθοδήγησε, μας ενέπνευσε για την επιλογή του θέματος, ιδίως ό,τι αφορά το επίπεδο φιλοδοξίας και το πολύ ευρύ πεδίο αυτής της στρατηγικής. Η αρχική μας ιδέα, για να είμαι και ειλικρινής, ήταν ε, μια στρατηγική για τις πτυχές ασφάλειας ε, στις θάλασσες, αλλά τελικά ε, οδηγηθήκαμε σε μια ευρύτερη προσέγγιση επαναλαμβάνω περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερα και λόγω του τρόπου με τον οποίο εργαστήκαμε, δηλαδή σε πολύ στενή συνεργασία και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσω, δεν ήταν απλά συντονισμός, ήταν μια κοινή εργασία. Υπήρξαν ε, σίγουρα κοινά προβλήματα, αλλά υπήρξε κοινή δουλειά και αυτό ήταν ε, άκρο θετικό εμπειρία για εμάς. Προσπαθήσαμε και τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν ε, στην προσπάθεια εντός βέβαια των ορίων της εκπόνησης μιας ε, ανακοίνωσης, επικοινωνίας μας, αλλά καταφέραμε, πιστεύω, να δώσουμε στα κράτη-μέλη και ένα αίσθημα ε, ιδιοποίηση αυτής της στρατηγικής. Και τώρα που έχουμε αυτή τη στρατηγική θα την ολοκληρώσουμε και η Ελληνική Προεδρία σε αυτή τη φάση καταρτήσει ένα μηχανισμό συντονισμού για να μπορέσουμε να έχουμε επίσημα ε, συμμετοχή από τα κράτη-μέλη. Πάντως, επειδή είχαμε διαβουλεύσει με τα κράτη-μέλη, από την αρχή είχαν συμμετοχή στις εργασίες μας. Κατά την άποψή μας, ε, ποιες είναι, χωρίς να επανέλθω ε, ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι ικανοποίησης για εμάς. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες. Ε, σας είπα ποιο είναι το γενικό πλαίσιο, ποια είναι η φιλοδοξία μας με αυτό το έγγραφο. Ο στόχος μας δεν είναι απλά να δούμε την ε, θαλάσσια ασφάλεια από το πρίσμα της ε, Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας. Πολύ γρήγορα διαπιστώσαμε ότι δεν θα έχει κανένα νόημα κάτι τέτοιο. και δεν το βγάλαμε από το μυαλό μας ε, σκεπτόμενοι απλά θεωρητικά, αλλά είναι ένα πρακτικό ε, συμπέρασμα που συναγάγαμε από την επιχείρηση Αταλάντη. Και επειδή είναι και άκρος ε, ποικίλα τα θέματα, μεταφορές, διαχείριση κρίσεων, περιβάλλον, τουρισμός, αλία και πάρα πολλά άλλα, Άρα πρέπει να τα εντάξουμε όλα αυτά τα θέματα σε μία ενιαία στρατηγική. Αυτό απαιτεί μία σφαιρική προσέγγιση. Υπάρχει όμως και μία ιδιαίτερη πτυχή στον τομέα της ασφάλειας. Εσωτερική ασφάλεια, εξωτερική ασφάλεια. Πώς διαρθρώνονται οι δύο πτυχές. Αυτό αποτέλεσε αντικείμενο πολλών συζητήσεων. Είχαμε πολλές συναντήσεις. Και αν υπάρχει ένας τομέας στον οποίο η διάκριση εσωτερικής ασφάλειας, εξωτερικής ασφάλειας πρέπει να εξαλειφθεί στη διαχωριστική γραμμή να σβήσει, είναι ακριβώς η ναυτική θαλάσσια ασφάλεια. Δηλαδή θα πούμε ότι σταματάει η Frontex ε, ε, εκεί που ξεκινά το γραμμή και όλα τα υπόλοιπα τα λαμβάνουν οι υπεύθυνοι για τις θάλασσες. Είναι Πολύ σοβαρά όλα αυτά τα θέματα πρέπει να μας απασχολήσουν. Δεύτερο ε, που μας ικανοποιεί είναι ότι καταφέραμε να βασιστούμε σε πρακτική εμπειρία για να αναπτύξουμε αυτή τη στρατηγική και για να ε, εντάξουμε τα διδάγματα που αντλήσαμε από τις επιχειρήσεις μας στο κέρας της Αφρικής. Ιδίω ό,τι αφορά την επιτυχία τη ασφάλεια. Και ιδίω μιλάω για την επιχείρηση Αταλάντη. Η επιχείρηση Αταλάντη, όπω γνωρίζετε, για πρώτη φορά στο Γενικό Στρατιωτικό Επιτελείο είχαμε εκπροσώπους της ναυτικής βιομηχανίας. Πάντοτε στο Γενικό Επιτελείο έχουμε έναν εκπρόσωπο της βιομηχανίας. Σε αυτή την επιχείρηση Αταλάντη αναπτύξαμε πάρα πολύ στενέ σχέσεις με μια σειρά άλλου φορεί, Διεθνή Αυτιλιακό Οργανισμό βέβαια, αλλά και τι επαγγελματικέ ε, ενώσεις, ε, τα ναυτικά επαγγέλματα. Αυτή η επιχείρηση ε, νομίζω πώς να το πω, ήταν ένα πιστικό επιχείρημα ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να αναλάβει την προεδρία της ομάδας επαφής για την πειρατεία από την Αγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Είμαστε λοιπόν εμείς που προεδρεύουμε φέτος αυτής της ομάδας επαφής. αυτή όλη η εμπειρία που συγκεντρώσαμε λοιπόν στο πλαίσιο αυτής της θαλάσσης στρατηγικής μας βοηθάει και αυτή η πολυμέρεια ακριβώς που εφαρμόζεται και στο πεδίο της ε, θαλάσσιας πολιτικής είναι κάτι που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε. Τρίτο ικανοποιητικό, ικανοποιητική, ικανοποιητική εξέλιξη είναι το ότι καταφέραμε να δημιουργήσουμε τα θεμέλια για διασύνδεση της δικής μας ευρωπαϊκής δράσης, αυτό που κάνουμε εμείς δηλαδή στον τομέα της ΕΠΑ και άλλες δράσεις, το τομέα της ανάπτυξης, άλλοι μηχανισμοί, άλλα μέσα. Πώς ε, συναρθρώνονται μεταξύ τους. Υπάρχουν προγράμματα, Μαρσίκ, Μαζέ, που δίνουν τη δυνατότητα στις χώρες της περιοχής να ελέγχουν καλύτερα το θαλάσσιο χώρο. Και αυτό το πρόγραμμα συμπληρώνει τις δικές μας δράσεις στο πλαίσιο της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Και με την Frontex συνεργαζόμαστε όλο και πιο στενά. Συνεργαστήκαμε όταν μαζί ε, αναλύσαμε την κατάσταση μετά την τραγωδία της Λαμπεντούζα και θέλουμε να συνεχίσει αυτή η συνεργασία. Για να ολοκληρώσω τώρα κύριε Πρόεδρε, όπως ε, προαναφέρθηκε, ναι μεν έχουμε πίσω από αυτό το έγγραφο πάρα πολλή δουλειά, αυτό είναι όμως η αφετηρία μας, δεν είναι η κατάληξη. Πρέπει να δώσουμε επιχειρησιακό χαρακτήρα σε αυτή τη στρατηγική τώρα. Γιατί τέλος δεν έχει νόημα. Η Κομισιόν έχει μακρά εμπειρία στο να δίνει επιχειρησιακό χαρακτήρα σε τέτοιου είδους έγγραφο. Πρέπει να δούμε τις επιτυχίες ε, της ασφάλειας, της κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας και πώς αυτή μπορεί η πολιτική να προσφέρει όλη της την προσθέμενη αξία, όλα τη τα μέσα και εργαλεία για να στηρίξει μια πραγματικά ευρωπαϊκή στρατηγική. Τι διδάγματα μπορούμε να αντιλήσουμε από την Αταλάντη στο τεφατό διάλογο και τη σχέση με τις ναυτικές, ε, ναυτιλιακές αρχές, πώς μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα το θέμα της ε, επιτήρησης των θαλασσών. Αυτά ε, διακυβεύονται στις επόμενες συζητήσεις. Αυτές είναι μελλοντικέ προκλήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω και εγώ μια ερώτηση. Όσον αφορά τον τρόπο που εσείς εστιάζεστε περισσότερο στο γεωγραφικό πεδίο, στο θέσουμε έτσι όσον αφορά τις θάλασσες, ε, τους ωκεανούς ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα. Βέβαια, ξέρουμε ότι ορισμένε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν και υπερπόντια εδάφη. Πάντω γνωρίζουμε πολύ καλά πώ λειτουργούν τα πράγματα για τη Μεσόγειο, τη Βαλτική κτλ. Πώ όμω μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια στη θάλασσα για τι υπόλοιπε θάλασσε, για του άλλου ωκεανού, για άλλε περιοχέ του κόσμου. Ξέρουμε τι, τι γίνεται, για παράδειγμα, για την καταπολέμηση πειρατεία στον Ινδικό ωκεανό ωστόσο υφίστανται κάποια ερωτήματα και κάποια ζητήματα ασφάλειας και εμπορικής ασφάλειας πολλές φορές σε άλλες περιοχές του κόσμου, σε κάποιους πολύ πιο μακρινούς ωκεανούς, όπου μόνο λίγα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελικά έχουν μια κάποια παρουσία από θαλάσσιας πλευράς όσον αφορά το ζήτημα της ασφάλειας. Αναφέρουμε για παράδειγμα στις χώρες της Ασίας, στην περιοχή της Ασίας. Πώς μπορούμε να καλύψουμε εμείς αυτό το γεωγραφικό πεδίο το εγκαταλείπουμε εντελώ, δεν ασχολούμαστε με αυτό, εφαρμόσουμε κάποιες γενικές αρχές ή μπορούμε τελικά να έχουμε μια πιο συγκεκριμένη δράση ευρωπαϊκή στην περιοχή αυτή, σε αυτούς τους μακρινούς ωκεανούς, στις μακρινές αυτές θάλασσες. Αυτή είναι η δικιά μου ερώτηση. Η κυρία Κοπά θέλει το λόγο. Φαντάζομαι εξ ονόματος της κυρίας Γκόμες επίσης, ε, κυρία Κοπά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Στα πλαίσια της Επιτροπής αυτής, το ζήτημα της ασφάλειας στη θάλασσα μας έχει απασχολήσει ιδιαιτέρως. Περιμέναμε τη δική σας την ανακοίνωση πριν την σύνοδο του Δεκεμβρίου. Επομένως την χαιρετίζουμε. Θα κάνω εγώ κάποιες παρατηρήσεις και συνέχεια θα αναφερθώ σε κάποια σχόλια της κυρίας Γκόμες. Πότε πιστεύετε ότι οι κρατών και κυβερνήσεων θα είναι σε θέση να εγκρίνουν τελικά το κείμενο. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς ευρωπαϊκές εκλογές, μπαίνουμε σε μια μεταβατική φάση όσον αφορά τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύετε ότι αυτό θα μας καθυστερήσει σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα το οποίο προβλέπετε. Εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε άμεσα να εγκρίνουμε τη στρατηγική αυτή και να αρχίζουμε να εργαζόμαστε βάσει αυτή τη στρατηγική. Αυτή είναι η δική μου ερώτηση, να διαβάσω τώρα την ερώτηση και τα σχόλια τη κυρία Γκόμε. Είχα τη δυνατότητα να διαβάσω την πρόταση, την ανακοίνωση μάλλον τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την ασφάλεια στη θάλασσα και θεωρώ ότι θα πρέπει πραγματικά να χαιρετήσουμε τις προτεραιότητες τις οποίες έχει εντοπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τον τομέα της ασφάλειας τη θάλασσα. Εγώ παρόλα αυτά βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες αδυναμίες. Σε καμία περίπτωση δεν βλέπουμε η κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα να έχει έντονο ρόλο όσον αφορά την μελλοντική στρατηγική για την ασφάλεια στη θάλασσα. Διακόπτει ο πρόεδρος. Σε καμία περίπτωση δεν βλέπουμε η κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα να έχει κεντρικό ρόλο όσον αφορά την μελλοντική στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια στη θάλασσα. Και όντω αυτό μπορεί να είναι επιζήμιο όσον αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη τη θάλασσια διάσταση τη κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα, αλλά είναι επιζήμιο επίση και τη δυνατότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να καταφέρει να αντιμετωπίσει όλου αυτού του κινδύνου η τι απειλέ, στην πολύ δυνητικού που εντοπιζονται στην ανακοινωση αυτη πολυ σωστα ομω η ανακοινωση από την EU-NAFOR και την επιχείρηση Αταλάντα και ότι όντω χρειάζεται ένας καλύτερος συντονισμός προκειμένου να κάνουμε αυτή τη στρατηγική και την αμυντική πτυχή της πιο αποτελεσματική. Η επιτυχία άλλωστε της επιχείρησης Ανταλάντα έχει να κάνει με το ότι είχαμε μια προσέγγιση sui generis και αποτελεί αυτό μοναδικό επίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια αποστολή, για μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί τόσο πολιτικά και στρατιωτικά μέσα η συνθήκη της Λισαβόνας στα πλαίσια της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ζητά μία περαιτέρω ανάπτυξη της πολιτικής αυτής. Οποιαδήποτε στρατηγική ασφάλεια στη θάλασσα θα πρέπει πραγματικά να βασίζεται στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας ανεξάρτητα από τους φορείς που εμπλέκονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ε, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στη θάλασσα θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στους στόχους της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Αυτό προσπάθησε να πετύχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μέσω της δικής μου έκθεσης για την θαλάσσια διάσταση της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας είναι να καταφέρει να εντοπίσει ε, στις δυνατότητες επιτυχούς στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στη θάλασσα μέσω της χρησιμοποίησης της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Τώρα, όσον αφορά το pooling and sharing, τον περισμό και την κοινή χρήση, γίνεται μία αναφορά στο κείμενο. παρόλα αυτά, δεν γίνεται κάποια στεναρή αναφορά στο κείμενο όσον αφορά την περαιτέρω χρησιμοποίηση τη μεθόδου pooling and sharing για κάποιε υποδομέ ε, ζωτική σημασία θεωρώ ότι το pooling and sharing μπορεί να αποτελέσει πολύ σημαντική πτυχή τη στρατηγική για την ασφάλεια στη θάλασσα, ιδίω στα πλαίσια τη ε, τρέχουσα οικονομική κρίση, όπου βλέπουμε ότι παντού στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια μείωση των αμυντικών ε, δαπανών. Όντω, ε, η πρωτοβουλία αυτή έχει προωθηθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα, αλλά έχει έρθει πλέον η κατάλληλη στιγμή για όλα τα κράτη-μέλη να συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορούν από μόνο τους να κινηθούν μόνο σε εθνικό επίπεδο. Αντίθετα, από κοινού, μέσω της κοινή συνεργασία μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα. Υπό το φω λοιπόν όλων αυτών είναι λυπηρό, αλλά δεν δηλαδή, μα προκαλεί έκπληξη, το ότι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αναφέρεται καθόλου στην εργασία που έχει επιτελέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το σημείο αυτό λήφθηκαν υπόψη από όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απόψει τη υποπιτροπή μα και πιστεύω ότι θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται και στην ανακοίνωση στρατηγική. Ω προ αυτό λοιπόν νομίζω ότι εκπροσωπώ την πλειοψηφία των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν καλό το, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δείξει ιδιαίτερη πυγμή και να χρησιμοποιήσει τελικά τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ανακοίνωσή τη. Δεν πρόκειται για ένα νομοθετικό ζήτημα, αυτό το γνωρίζουμε, αλλά παρόλα αυτά αισθάνομαι μια κάποια μηχανία όταν βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλο και πιο συχνά δεν λαμβάνει υπόψη τη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν δεν συζητούμε ζητήματα συναπόφαση. Εκπροσωπούμε εμεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Ευρωπαίου πολίτε, για αυτού εργάστε και εσεί και θεωρώ ότι στο όνομα των Ευρωπαίων πολιτών θα πρέπει να αναπτύξουμε μια καλύτερη πολιτική για την ασφάλεια στη θάλασσα. Του των θα ήθελα να χαιρετήσω για άλλη μια φορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι στη σωστή κατεύθυνση, μόνο ότι θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας πιο έντονος ρόλος για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, καθώς επίσης και για την ύπατη εκπρόσωπο, η οποία είναι και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μόνο μια στεναρή ισχυρή στρατηγική πολυτομιακή, η οποία θα βασίζεται σε συντονισμό, σε πολλά και διάφορα επίπεδα, μόνο μια στρατηγική η οποία θα είναι οικονομικά αποδοτική και που θα τυχαίνει ευρωπαϊκή διαχείριση, μόνο μια τέτοια στρατηγική θα είναι τελικά επιτυχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να εγκρίνουμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια στη θάλασσα και μέσω αυτή να καταφέρουμε να επιλύσουμε και διάφορα προβλήματα θεσμική συνεργασία που αντιμετωπίσαμε στο παρελθόν. Βλέπω ότι η είτε μιλάει είτε γράφει είναι πάντα πάντα μέσα στα πράγματα. Πάντα, πάντως είναι πάρα πολύ εξονυχιστικό αυτό το οποίο έχει γράψει και η έκθεσή της φυσικά είναι πάρα πολύ φιλόδοξη. Είναι απόλυτα λοιπόν λογικό να τονίζει τα επιχειρήματά της. <clears throat> κυρία Μίντερ και κύριε Λενουάρα αν θέλετε. Α, συγγνώμη, ο κύριος Γιάννης θέλει να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ίσως θα θέλουν οι καλεσμένοι μας να απαντήσουν πρώτα στην κυρία Κοπά. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αν μπορώ να λάβω τώρα το λόγο, θα έλεγα το εξή. Θέλω με συντομία να εστιάσω στο εξή θέμα. Όταν άκουσα τις παρεμβάσεις σας, σκεφτόμουν, όπως κάνουμε πάντα ως πολιτικοί, τον απλό πολίτη, για τον οποίο εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Δεν ξέρω λοιπόν αυτά τα 500 εκατομμύρια πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν μπορούν να καταλάβουν κάτι το οποίο για μένα φαίνεται υπερβολικά τεχνικό και γραφειοκρατικό. Δεν νομίζω ότι μπορούν να καταλάβουν εύκολα οι πολίτες μας ακριβώς γιατί μιλάμε σήμερα. για την ε, στρατηγική λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει η, στρατηγική, η κοινή στρατηγική που είχε διατυπώσει ο Χαβιέ Σολάνα το 2003. Αυτό είναι το προηγούμενό τη αν θέλετε, της σημερινής αυτής πρότασης. Και η οποία πέρασε από 40 κύματα στο παρελθόν. Και τώρα ουσιαστικά δημιουργείται και πάλι από την αρχή. Η Επιτροπή μας λοιπόν έχει αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα και συζητήσαμε για να μπορέσουμε να διακριβώσουμε ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες ασφάλειας και αντίθετα οι παράγοντες απειλής κατά της ασφάλειας της Ευρώπης και με ποιο τρόπο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις δυνητικές ε, απειλές. Όλα αυτά όμως είναι τόσο ευ είναι τόσο ευρία αυτή η αντιμετώπιση που αντιμετωπίζει από τα κράτη που έχουν αστοχήσει μέχρι τη διεθνή τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. Όλα αυτά είναι θέματα που έχουμε αντιμετωπίσει με μεγάλο ενδιαφέρον σε προηγούμενες θητείες. Αλλά αυτό το έγγραφο το οποίο βλέπω να συνοδεύει τη δική σας παρουσία εδώ δεν βλέπω να αναφέρεται καθόλου στα πρόσφατα γεγονότα της Κρυμαίας και στην Μαύρη Θάλασσα. Η Μαύρη Θάλασσα είναι μια περιοχή μεγάλης στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί βρέχονται από τη Μαύρη Θάλασσα διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι φυσικά εκεί που περνάει, είναι ο χώρος από τον οποίο περνάει ο Σοβιετικός στο παρελθόν, η Ρωσικός στόλος, τώρα στην Μεσόγειο. Πέραν λοιπόν πέραν το, της ιστορικής σημασίας που μπορεί να έχει ο πόλεμος Κρυμαίας το 1850 τόσα και που μπορεί να έχει παρόμοιες αιτίες με το σημερινό, έχουν αλλάξει φυσικά τα τεχνολογικά δεδομένα και στρατιωτικά δεδομένα, παραμένουν ορισμένοι παράγοντες οι οποίοι είναι πάγοι Η στάση της Ρωσίας είτε είναι αυτοκρατορία είτε δεν είναι αυτοκρατορία, είτε είναι ένα κράτος το οποίο είναι αυτοκρατορικό είτε είναι ένα κράτος δικτατορικό Λοιπόν, ανεξάρτητα από τη μορφή που έχει η Ρωσία σε όλες αυτές τις χρονικές στιγμές, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι που τουλάχιστον ο πληθυσμός ορισμένων χωρών τις αντιμετωπίζει ως γεωγραφικά πολύ κοντινές του. Και επίσης διαπιστώνει ή αντιλαμβάνεται τουλάχιστον μια ηγεμονική ή επεκτατική διάθεση από την πλευρά της ε, Ρωσίας του Πούτιν. Θα ήθελα λοιπόν να θέσω το ερώτημα και αυτό είναι ένα ερώτημα για τους υπουργούς των κρατών που εμπλέκονται στο θέμα αυτό περισσότερο και είναι ερώτημα προς την υψηλή εκπρόσωπο, μήπως θα είχε νόημα να αντιμετωπίσουμε καλύτερα το θέμα αυτό και επίσης η πολιτική αποστολή που έχουμε στείλει στη Γεωργία έχει ένα αντικείμενο ε, παρόμοιο που είναι η αντιπαράθεση μεταξύ του κράτους της Γεωργίας και της Ρωσίας για ορισμένε εδαφικές περιοχές της Γεωργίας. Όλα αυτά λοιπόν με φέρνουν να υπενθυμίσω σε κάτι το οποίο έλεγε ο πρόεδρος Πούτιν και το έχει πει κατά, κατά επανάληψη ότι όπου υπάρχουν Ρώσοι Ρώσοι υπήκοοι, όχι Ρώσοι υπήκοοι, αλλά Ρώσοι εθνοτικοί ε, στις χώρες αυτές, η Ρωσία έχει την υποχρέωση και το καθήκον να τους υπερασπιστεί. Έχουν περάσει λοιπόν έξι χρόνια σχεδόν από το 2008 και κατά τη δική μου άποψη σε πολιτικό, σε στρατιωτικό, σε σχεδιαστικό και στρατηγικό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει προχωρήσει σχεδόν καθόλου ούτε σε επίπεδο συνεργασίας με τη Ρωσία για να αποτραπεί η επανάληψη τέτοιων γεγονότων ή τουλάχιστον να μπορούν να προβλεφθούν εκ των προτέρων και να ενεργοποιηθούν μηχανισμοί για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Ούτε από την άλλη πλευρά έχουμε ακολουθήσει μια στρατηγική που να πούμε ότι η Ρωσία είναι ένας αντίπαλος, είναι ένας ανταγωνιστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια δύναμη με την οποία εμείς θα πρέπει να έχουμε μια ε, σωστή αντιμετώπιση. Βλέπετε το πρόβλημα τώρα της Κρυμαίας και της Ουκρανίας. Πρέπει, αν η Ουκρανία θέλει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, εμείς να διαβουλευτούμε πρώτα με τη Ρωσία ή θεωρούμε ότι η Ουκρανία έχει την εθνική της κυριαρχία. Όλα αυτά είναι τα ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί και είναι ζωντανά ακόμα στον, στο Συμβούλιο των Υπουργών, στην Κομισιόν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γενικά στην κοινή γνώμη της Ευρώπης. Λοιπόν, πρέπει εφόσον μιλάμε για μια θαλάσσια στρατηγική, να λάβουμε υπόψη όχι μόνο τη Μεσόγειο, αλλά και την ε, Μαύρη Θάλασσα. Και δεν άκουσα τίποτα για τη Μαύρη Θάλασσα που είναι κάτι που συνδέεται ιδιαίτερα με την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη δική μου άποψη είναι το πιο σημαντικό ζήτημα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα στην Ευρώπη. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να έχουμε και κάποιες κατευθύνσεις για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά που εγείρονται στη Μαύρη Θάλασσα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω περισσότερο. Απλώς ήθελα να θέσω αυτά τα ερωτήματα. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα δώσω στους δύο μιλητές μας το λόγο. Η κυρία Γκνίντερ πρώτα. Ευχαριστώ πολύ, πολύ για τις ερωτήσεις σας. Πρέπει να σας πω ότι σίγουρα για το, τα περί της ε, κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας θα επεκταθεί πιο πολύ ο κύριος Λενουά. Στόχος μας βέβαια είναι να ξεπεράσουμε ε, αυτό το πεδίο και μας το Τήσε και η κυρία Κόμη στην έκθεση. Δεν ήταν και ο πιο εύκολος στόχος αυτός, γιατί και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου προέρχονται από αυτή την ε, πολιτική και έγινε και μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσον αυτό είναι ένα κομμάτι της ε, στρατηγικής. Και έπρεπε να πάρουμε και τη συμφωνή γνώμη των ε, εθνικών κυβερνήσεων. Πώς λοιπόν μπορούμε να τα εξισορροπήσουμε όλα αυτά. Αυτό μας απασχόλησε. Νομίζω ότι το καταφέραμε. Προσπαθώντας να έχουμε βέβαια ένα συμβιβασμό. Για τη συνεργασία με το Συμβουλίο σίγουρα θα επανέλθει το θέμα. Μας ενδιαφέρει και η δική σας συμβολή, οι δικές σας απόψεις. Σίγουρα είναι το χρονοδιάγραμμά μας φιλόδοξο. Ήδη συνεδριάσαμε δύο φορές ε, στο Συμβούλιο σε διάφορους σχηματισμούς. Τώρα ξεκινάει η δουλειά. Οπότε περιμένουμε έγκριση από τους αρχηγούς καρτών και κυβερνήσεων. Περιμένουμε με την Ελληνική Προεδρία να έχουμε ολοκληρώσει, δηλαδή μέχρι τις 26 Ιουνίου που συνεδριάζει το Συμβούλιο και η στρατηγική βέβαια από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Αλλά ελπίζουμε στα συμπεράσματα οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων να κάνουν θετική μνήα στη στρατηγική αυτή. Και έπειτα ξεκινά, όπως είπα, η πραγματική δουλειά με την ελοποίηση, την εφαρμογή και εκεί πιστεύω ότι μπορούμε να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες και επίσης να συμπεριλάβουμε και τις αναλυτικές απόψεις όλων των φορέων και του Κοινοβουλίου. Διαβάζοντας όμως την έκθεση Γκόμες και όταν ήταν ακόμα σε σχέση, στη φάση του σχεδιασμού, είχα πολύ ικανοποιηθεί γιατί είδα ότι είχε πολλές από τις ε, ιδέες μας αυτή η έκθεση. Και το βλέπω βέβαια και στην τελική έκθεση. Λαμβάνουμε υπόψη λοιπόν το input δική σας ε, επιτροπή. Η συγκέντρωση και η χρήση πόρων, pooling and sharing θα τα πει ο Didier. Πάντως είμαστε και εμείς δεσμευμένοι και προσιλωμένοι σε αυτή την αρχή. Πόσο γενναίοι και τολμηροί μπορούμε να είμαστε και τι κάνουμε ακριβώς αυτό θα εξαρτηθεί, ξέρετε, από όλους ε, τους άλλους παράγοντες, όχι μόνο από την Κομισιόν. Εμείς όμως στην Κομισιόν είμαστε αποφασισμένοι να πετύχει, ε, να εγκριθεί η στρατηγική. Και σχετίζεται και με αυτό που ο κύριος Γιάννης. Ήδη έχουμε επιτεύγματα, δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Και αυτό πρέπει να το μεταδώσουμε στους πολίτες μας. Υπάρχει προστασία, υπάρχει νομοθεσία, υπάρχουν φορείς, υπηρεσίες και συνεργαζόμαστε ενεργά με αυτούς τους οργανισμούς. Σίγουρα μπορούμε να βελτιωθούμε, αυτό λέμε και αυτό μπορούμε να το κάνουμε σε μια σχέση εταιρική με αυτό τον προσανατολισμό, γιατί μπορούμε να ωφεληθούμε από τη διαθεσιμότητα στρατιωτικών μέσων και μη στρατιωτικών μέσων που πρέπει να συνεργάζονται ο στρατιωτικός και μη στρατιωτικό τομέας, να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν στον δυνατόν καλύτερα τα μέσα και τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους. Δέχομαι λοιπόν ότι μπορεί να ακούγεται άκρο τεχνικό, αλλά έχει και πολύ σημαντικέ επιπτώσεις για τους πολίτες με όλο αυτό. Αν μιλάει κανεί για διαλειτουργικότητα, μεταξύ συστημάτων, μεταξύ αεροσκαφών, πλοίων. Ξέρετε, η επικοινωνία δεν είναι κάτι αυτόματο, δεν υπάρχει ένα διαδίκτυο. Άρα εδώ μπορούμε να κερδίσουμε σε θέματα απόδοσης σπόρων. Θέλουμε να υπάρχει μια πραγματική εταιρική σχέση μεταξύ αρχών που μέχρι στιγμής δεν συνεργάζονται πραγματικά μεταξύ τους και αυτό είναι το κλειδί για να έχουμε την έγκαιρη αντίδραση όταν αυτό απαιτείται σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και ακριβώς αυτό μπορούμε να το προσφέρουμε και για την περιοχή της Κρυμαίας. Φυσικά και δεν σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να αντιδρούμε αμέσως με αυτή τη στρατηγική, αλλά υπάρχει πλέον η βάση, υπάρχουν τα θεμέλια για να έχουμε μια καλή συνεργασία. Σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί, επαναλαμβάνω. Για το γεωγραφικό πεδίο, ίσως ο Ντιτιέ να πάρει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Για το γεωγραφικό πεδίο και εύρος, η θαλάσσια ναυτιλιακή αυτή στρατηγική από μόνη της δεν μπορεί κατά ανάγκη να δώσει από μόνη μια απάντηση σε αυτό το θέμα της γεωγραφικής κάλυψης που θα πρέπει να οριστεί όπως υπογραμμίστηκε στο πλαίσιο τους γενικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα ορίζει και τις προνομιακές ε, περιοχές δράσης εφόσον θα ορίζει και τους στόχους. Για τον τομέα της ασφάλειας, μας το λέει και επικαιρότητα σήμερα, πού είναι ακριβώς αυτές οι περιοχές κέρας Αφρικής, ο κόλπος της Γουινέας, ίσως Ασία, Νοτιοανατολική Ασία, για την ασφάλεια του εφοδιασμού μας, επιτήρηση ίσως άλλων στρατηγικών περιοχών, η στρατηγική διέλευση, έξινος πόντος, Μεσόγειος θα έλεγα εγώ, το έδειξαν και τα γεγονότα της περσινής χρονιάς, πόσο μεγάλη σημασία έχει η περιοχή της Μεσογείου. Άρα, σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κάλυψη, νομίζω ότι η απάντηση θα δοθεί μαζί με την αναγνώριση των ε, βασικών ευρωπαϊκών στόχων και όχι ε, απαραίτητα στο πλαίσιο της θαλάσσιας στρατηγικής που υπάρχει μεν, και υπάρχει για να αποτελέσει ένα επιπλέον εργαλείο που θα δώσει τη δυνατότητα εν συνεχεία σε όλους μας να μπορέσουμε να περιφρουρήσουμε και να προσπίσουμε τα συμφέροντά μας. Σε ό,τι αφορά το ρόλο της κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας, ερώτηση Γκόμες, αν θα πρέπει δηλαδή να έχει έναν κομβικό ρόλο. Δεν είμαι πεπισμένος ότι αυτή η πολιτική πρέπει να έχει ένα κομβικό ρόλο στη θαλάσσια στρατηγική. Πιστεύω ότι πρέπει να τη δούμε σε συνάρτηση με άλλες πολιτικές και μέσα, όπως είναι η Frontex, μέσω στήριξης πολιτικής, ή έλεγχος αλίας κτλ. Όταν έχουμε ένα πρόβλημα συγκεκριμένο, ad hoc, κατά περίπτωση, θα διαρωτούμαστε για το ποιο είναι το μείγμα πολιτικής που θα πρέπει να εφαρμόσουμε για να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά το εκάστοτε πρόβλημα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ανεξαρτήτω του προβλήματο θα πρέπει να έχει κομβικό ρόλο η κοινή πολιτική άμυνα και ασφάλεια, γιατί μου φαίνεται ότι αυτό θα μα οδηγήσει σε πάρα πολύ βιαστικά συμπεράσματα. Ενώ θα μπορούσαμε ενδεχομένω να εξετάσουμε άλλε απαντήσει, ανάλογα με το κάθε πρόβλημα, παραλαμβάνω. Το policy mix αποφασίστηκε την εντόπιση ενό δεδομένου προβλήματο, γιατί περί αυτού πρόκειται. Να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένε ε, περιπτώσει, κόλπο Γουινέας, έλεγχος ε, της Ανατολικής Μεσογείου, ασφάλεια φοδιασμού ε, στον κόλπο της ε, Μαλάκα κτλ. Εκεί αποφασίζεται κατά περίπτωση με ανάλυση διεξοδική σε βάθος που είναι τα συμφέροντά μας, τι προβλήματα μπορεί να ανακύψουν, ποιους, ποιοι είναι οι λόγοι τους οποίους δεν έχουν ρυθμιστεί τα προβλήματα από αυτούς που θα έπρεπε να το επιλύσουν τα προβλήματα, τα προβλήματα αυτά και από και τα ορίσουμε όλα αυτά μπορούμε να χαράξουμε την ε, στρατηγική μας για μια παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το ρόλο λοιπόν της ε, και ΠΑ, πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι ευέλικτο ο ρόλο και να προσαρμόζεται στι ιδιαίτερε συνθήκε και περιστάσει, ανάλογα με την περίπτωση δηλαδή. Για την παρουσίαση αυτή τη ε, θαλάσσια στρατηγική στου Ευρωπαίου πολίτε. Όλο το θέμα είναι επιχειρησιακό χαρακτήρα χαρακτήρας που θα δοθεί σε αυτή τη στρατηγική. Δεν είναι εύκολο να παρουσιάσει κανεί αυτό το τόσο θεωρητικό κείμενο στου Ευρωπαίου πολίτε. Πολύ πιο εύκολο μπορεί να πλασάρει εντό αγωγικών την πρακτική του εφαρμογή, την επιχειρησιακή του πτυχή. Και αυτό θα είναι και το αντικείμενο των μελλοντικών μα συζητήσεων. Η στρατηγική, επομένω, σίγουρα δεν μπορεί να παραμεριστεί, γιατί θα είναι η βάση, είναι να αναπόσπαστο τμήμα αυτής της διαδικασίας, αναγκαίο, εκ των όνου κάνευ, αλλά δεν είναι το μόνο. Θα πρέπει να πούμε δε στους πολίτες ότι ορίστε αυτή η θαλάσσια στρατηγική είναι η βάση ε, πάνω στην οποία θα αποφασίζονται οι μελλοντικέ δράσεις. Ή αποφασίζονται κάποιες δράσεις και μπορούμε να δώσουμε παραδείγματα. Αυτά είχα να πω, δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι. Σας ευχαριστούμε. Θέλω να ξαναπάρουν το λόγο συνάδελφοι μετά τις εξηγήσεις μας έδωσε ο κύριος Λενουάρ. Αν όχι, τότε σας ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν την επίσημη αυτή ε, ανακοίνωση και προφανώς το ζήτημα αυτό θα μας απασχολήσει και στο μέλλον και όσον αφορά όλες τις υπόλοιπες στρατηγικές, τις οποίες ξεχάσαμε σήμερα, Πιστεύω ότι ε, το επόμενο κοινοβούλιο θα ενδιαφερθεί ιδιαίτερα και για την εφαρμογή τους. Γιατί δυστυχώς στο παρελθόν είδαμε ότι υπήρχαν πολύ καλές ε, στρατηγικές από θεωρητικής πλευράς, η παρουσίασή τους ήταν τέλεια, αλλά στην πράξη είδαμε ότι ε, η εφαρμογή τους δεν ήταν ικανοποιητική. Νομίζω λοιπόν ότι Πολλές φορές με διάφορες στρατηγικές όπως και στο Σαχέλ είδαμε ότι χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια για να καταφέρουμε τελικά να ελοπίσουμε αποτελεσματικά την ελόγω στρατηγική στην πράξη. Σας ευχαριστούμε πάντως πολύ. Καλή συνέχεια. Θα κάνουμε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα περιμένοντας τον ε, υποπτέραχο Βαλεντά. Κύριε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε σας παρακαλώ. Σα το συγγνώμη για το σύντομο αυτό διάλειμμα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έχουμε ανάμεσά μας σήμερα τον υποπτέραχο Βαλεντά, ο οποίος είναι επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Επιτελείου Ενερίων Μεταφορών στο Αϊντόβεν των Κάτω Χωρών, γνωστό και ω EUATC, ε, EATC μάλλον με συγχωρείτε, πριν από 1,5 χρόνο ήταν εδώ ο προκατοχός σας, ο οποίος μας είπε και το βλέπουμε ότι πραγματικά μιλάμε για ένα success story, μια ιδιαίτερη επιτυχημένη ιστορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χαιρόμαστε λοιπόν πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα μαζί μας, επιτυχημένο το όλο εγχείρημα, διότι η δομή αυτή λειτουργεί πολύ καλά και επειδή από πολιτικής πλευράς Πρόκειται για ένα παράδειγμα το οποίο πραγματικά μας εμπνέει. Και το βλέπουμε αυτό στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, όπου αναφερόμενο σε ζητήματα άμυνας, και σας λέω κύριε Υποπτήραρχε ότι εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε υποβάλει κάποιες επικρίσεις, είχαμε εκφράσει μάλλον την απογοήτευσή μας σχετικά με τις φιλοδοξίες που εξέφρασε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την έλλειψη μάλλον φιλοδοξιών. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι υπήρχαν κάποια πολύ θετικά συμπεράσματα όσον αφορά το EATC. Αναφερόταν ε, το έγγραφο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο πολύ θετικό έργο, τα πολύ θετικά αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Επιτελείου Νερίου Μεταφορών, αλλά και στην επικείμενη διεύρυνσή του, καθότι η Ισπανία πρόκειται να προσχωρήσει στο EATC. Οι αρχηγοί πάντως κρατών κυβερνήσεων είπαν επίσης ότι πέρα από τη διάρθρωση και τη δομή του EATC, το EATC αποτελεί και ένα πολύ θετικό παράδειγμα συνεκμετάλλευσης και επιμερισμού. Ας μην ξεχνάμε ότι το EATC δεν αποτελεί δομή όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόκειται απλώς για έναν θεσμό ευρωπαϊκής συνεργασίας ανάμεσα σε κράτη-μέλη τα οποία οικειοθελώς συμμετέχουν. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπενθυμίσουμε το εξή, πράγμα το οποίο μα ενδιαφέρει και εμά ιδιαίτερα όσον αφορά τη λειτουργία του, είναι ότι το Ευρωπαϊκό Επιτελείο Ενεργείων Μεταφορών σε καμία περίπτωση δεν υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να αποποιηθούν την κυριαρχία του όσον αφορά τι εθνικέ του ικανότητε. Ουσιαστικά τα κράτη-μέλη εκχωρούν την υποδομή τους, τα μέσα τους τον εξοπλισμό τους μάλλον, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευση, συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μια βελτιστοποίηση των πόρων σε ένα τομέα ο οποίο είναι θεμελιώδου σημασία όσον αφορά τις ε, ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνατότητες. Επιμένω πάντως σε αυτόν τον καινοτόμο χαρακτήρα του ε, EATC το, και θα μπορούσε ο χαρακτήρας αυτός να αποτελέσει και να επιπλέον μοντέλο στρατιωτικής συνεργασίας και για άλλους τομείς, δηλαδή ότι τα κράτη-μέλη διατηρούν την ιδιοκτησία, την κυριαρχία των στρατικών τους μέσων και απλώς επιτρέπουν την, να αποτελέσουν αντικείμενο συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι το μοντέλο αυτό ανταποκρίνεται πραγματικά σε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και σε άλλους τομείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια. Κάθε φορά προσπαθούμε να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο. Δεν είμαι εγώ υπέρ μια τέτοια προσέγγιση. Ορισμένοι πάντω θέλουν να έχουμε μια συνολική σφαιρική συνεκμετάλλευση των στρατιωτικών μέσων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν λοιπόν να προχωρήσουμε στην κατεύθυνση αυτή, νομίζω ότι μπορούμε να βασιστούμε στην εμπειρία του Ευρωπαϊκού Επιτελείου Εναερίων Μεταφορών να δούμε επίσης και ποια είναι τα πλεονεκτήματα για τα κράτη-μέλη τα οποία συνεισφέρουν και για τα κράτη-μέλη τα οποία χρησιμοποιούν τα μέσα αυτά. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά κύριε Υποπτέραρχε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε στην Επιτροπή μας. Νομίζω ότι θα προβληθούν και κάποιες διαφάνειες. Γι' αυτό μειώνουμε και λίγο το φωτισμό στην αίθουσα. Έχετε ευθύς αμέσως το λόγο. και κύριοι, θα πω δύο λόγια στα γαλλικά μονάχα για να ευχαριστήσω τον ε, πρόεδρο τον Ζω για την πρόσκληση που μου απίθυνε και ο στόχος μας να σας κάνουμε μια επισκόπηση της κατάστασης της Ευρωπαϊκής Διοίκησης Εναερίων Μεταφορών, μεταφορών καλύτερα, και τα θέματα, να παρουσιάσω θέματα τα οποία θα σας ενδιαφέρουν. Έχω μαζί μου το συνταγματάρχη ε, Αλμπέρτο Μέντες, το Σμίναρχο Αλμπέρτο Μέντες που είναι από την Ισπανική, από την Ισπανική αεροπορία και τον ε, Σμίναρχο Βεριέ, ο οποίος είναι εκπρόσωπος των γαλλικών δυνάμεων μέσα στην Νέα Και έχουμε και ένα ε, μαθητευόμενο από την Πούδου ο, ο οποίος κάνει μαθητεία στην ε, ε και τώρα χωρίς καμία μετάβαση θα ήθελα να περάσω στα αγγλικά. Και θα ήθελα να σας πω ότι δυστυχώς αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα το καταδεικνύει οι εποχές, της, οι εποχές κρίσεων δεν πάβουν να υπάρχουν, θα συνεχίσουν και στο μέλλον. Ακόμα και αν οι προϋπολογισμοί μειώνονται, ελπίζω να διαψευστώ το πρώτο μου μήνυμα λοιπόν σε εσά είναι η συνεργασία λοιπόν δεν είναι πια επιλογή, είναι μια αναγκαιότητα. Σήμερα περισσότερο παρά ποτέ. Θα ήθελα να αφήσω το μέγιστο δυνατό χρόνο για ερωτήσεις και απαντήσεις. Θέλω να σας δείξω καταρχήν γιατί εμείς είμαστε ένα επιτυχημένο παράδειγμα του λεγόμενου pooling and sharing, της θέσης από κοινού και του διαμοιρασμού πόρων στην Ευρώπη. Έχουμε και μερικά αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν και τα οποία είναι πάρα πολύ θετικά, δηλαδή δημιουργούμε ένα αίσθημα εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης και επίσης συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της κοινή ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και φυσικά δεν είμαστε τέλειοι, δεν ζούμε σε ένα τέλειο κόσμο. Έχουμε και τις προκλήσεις ενώπιόν μας. Ε... Συγγνώμη για τις διαφορές αν υπάρχουν στα κείμενα. Η αποστολή μας είναι εξ των πέντε μελών της EATC, το Βέλγιο, η Γερμανία, οι κατοχώρες Λουξεμβούργο και η Γαλλία και αύριο ίσως η Ισπανία και το 2015 η Ιταλία, προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των ε, πόρων που έχουμε για αερομεταφορές και που έχουν αφοσιωθεί στην EATC. Αυτή είναι η καθημερινή μας ε, εργασία και θα επανέλθω στο σημείο αυτό αμέσως. Καταρχήν λοιπόν, έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική αντιμετώπιση. Είναι απλώς το γεγονός ότι σε καθημερινή βάση αντιμετωπίζουμε αποστολές, αποστολές αερομεταφορών για τις πέντε χώρες οι οποίες συμμετέχουν, ενώ συγχρόνως προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των μελών μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξηγήσω ότι αυτό είναι μια βασική αρχή. Αν θέλουμε να έχουμε καλή συνεργασία, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αποστολή, αν έχουμε λοιπόν μια αποτελεσματική λειτουργία, πρέπει να βελτιώνεται η ικανότητα συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων. Πρέπει λοιπόν να επιτευχθούν ορισμένοι στόχοι εναρμόνισης και τυποποίησης. Ο στόχος μας είναι φυσικά να εκτελέσουμε αποστολές για τα κράτη-μέλη μας και συγχρόνως να βελτιώσουμε την καλή τους συνεργασία. Αυτή είναι λοιπόν η βασική μας αντιμετώπιση και αντίληψη της αποστολής μας. Όπως είπε ο κ. Σταουζόν, αν θέλετε να συνεργαστείτε, αν θέλετε να κάνετε κάτι, θα πρέπει να μάθετε να διαβιβάζετε και κάποιες αρμοδιότητες, στη δική μας περίπτωση στην EATC. Αν δεν θέλει κανείς να μεταφέρει αρμοδιότητες, δεν θα μπορεί να συμμερίζεται πόρους και να τους θέτει από κοινού. Θα παραμείνει μονάχα μέσα στα στενά εθνικά πλαίσια. Σε πιο συγκεκριμένο λοιπόν επίπεδο μιλάμε για ένα δυνητικό στόλο περίπου 200 αεροσκαφών. Με την Ισπανία και την Ιταλία θα αυξηθεί βέβαια αυτός ο αριθμός αεροσκαφών. Και αυτό που είναι σημαντικό να καταγράψουμε είναι ότι αν θέλει κανείς να βελτιστοποιήσει τη χρήση αυτών των, των πόρων που είναι ουσιαστικά πόροι αερομεταφοράς, η επιτυχία εδώ εξαρτάται με την σωστή χρησιμοποίηση της εμβέλειας των πόρων αυτών. Και αυτό είναι ακριβώ αυτό που κάνουμε στο EATC, γιατί χρησιμοποιούμε αεροπλάνα όπως είναι τα ε, από DC-10 μέχρι Α340 ε, και αεροσκάφη κάσα σε 235 κτλ. Έχουμε 170 άτομα προσωπικό στη βάση του Eindhoven και από πέντε χώρες όπως είπα και θα φτάσουμε περίπου τους 200 όταν έρθει η Ισπανία και η Ιταλία. Πώς λειτουργούμε λοιπόν, τι κάνουμε στο Eindhoven. Τα αεροσκάφη μας φυσικά δεν βρίσκονται στο Eindhoven. Αυτό που κάνουμε είναι μας δίνουν κάποιους πόρους αεροσκάφη, δηλαδή τα κράτη-μέλη, και συγχρόνω μα ζητούν να εκτελέσουμε ορισμένες αιτήσει μεταφορών. Αυτό που κάνουμε λοιπόν, και αυτή είναι η αρχή του pooling and sharing, κάνουμε όσο μπορούμε περισσότερες αποστολές με τους σπόρους που έχουμε. Χρησιμοποιούμε λοιπόν αυτούς τους σπόρους ε, ανεξάρτητα από ποιο κράτος προέρχονται για να εκτελέσουμε αυτές τις αποστολές. Κάνουμε καταρχήν την αρχική σχεδίαση μιας αποστολής από το Eindhoven μαζί με τα κρατη περίπου έξι εβδομάδες πριν από την αποστολή και μετά έχουμε μια διαδικασία η οποία καταλήγει στην εκκίνηση της ε, αποστολής στέλνονται οι εντολές από το Άιντχόβεν στα πληρώματα των αεροσκάφων και οποιαδήποτε προβλήματα τα αναφέρουν όχι μόνο στα κράτη-μέλη τους αλλά και στο Άιντχόβεν ώστε να μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα της αποστολής. Γι' αυτό έχουμε αυτή την ε, διοίκηση αερομεταφορών γιατί έχουμε ακριβώς αυτές τις εξουσίες που έχουν διαδιδαστεί σε εμάς. Δεν θα πω πάρα πολλά <clears throat> για το τι έχουμε πετύχει στον λειτουργικό τομέα. Απλώς με αυτό το γράφημα σας δείχνει ότι το 2010 δημιουργηθήκαμε και ήμασταν πέρσι στο τέλος του περσινού χρόνου ήμασταν πλήρως λειτουργικοί και μάλιστα τα στοιχεία αυτά από το 2011 μέχρι το 2013 βλέπετε ότι τα αεροσκάφη που έχουμε στη διάθεσή μας έχουν μειωθεί κατά 30% από 66 την ημέρα σε 47 την ημέρα. Το, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι γυράσκουν οι στόλοι αλλά παρά το γεγονός ότι έχουν μειωθεί τα αεροσκάφη μας, έχουμε καταφέρει να διατηρήσουμε και τις μεταφορές φορτίων και τις μεταφορές επιβατών σε ένα επίπεδο που δεν ποικίλει παρά μόνο κατά 5% από το 2011. Αυτό είναι η βελτιστοποίηση. Με λιγότερος πώς μπορείτε να διατηρήσετε το ίδιο τελικό αποτέλεσμα. Δεν θέλω λοιπόν να σας δώσω πάρα πολλά στοιχεία, αλλά είναι εύγλωτο αυτό για να σας καταδείξει πώς εμείς μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τις αερομεταφορές. Σας είπα προηγουμένως ότι για να μπορεί κανείς να λειτουργήσει από κοινού πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση. Αυτό φαίνεται τεχνικό αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Χρειάστηκε να αλλάξουμε τους εθνικούς κανονισμούς για την ε, χρήση αεροσκαφών από την EATC. Αυτό αφορά πραγματικά χάρη τους κανόνες για την ε, για τις ώρες πτήσης, τις συνθήκες πτήσης, πόσες ώρες πρέπει να πετάξουν και πόσες ώρες πρέπει να ξεκουραστούν. Κάθε κράτος έχει τους δικούς του κανόνες και μπορέσαμε με τη βοήθεια αυτών των κρατών να δημιουργήσουμε ένα κοινό ε, αριθμό κανονισμών ώστε να χρησιμοποιούμε τα αεροσκάφη αυτά όσο πιο αποτελεσματικά μπορούμε. Ε, κοινή παροχή διπλωματικών αδειών έχουμε εξασφαλίσει με τα πέντε χρόνια κοινούς κανόνες για να δίδεται η, η άδεια υπέρπτυση με, πάνω από τι χώρε μα. Όλα αυτά μπορεί να φαίνονται πολύ εύκολα και προφανή, αλλά αυτό ήταν κάτι το οποίο μας κλείτωσε ε, πολύ χρόνο και εργασία. Και αυτό επετέφθη πάλι γιατί υπήρχε η θέληση συνεργασία. Επίση, προσπαθούμε να εναρμονίσουμε τις, ε, τα τακτικά προσόντα των ε, πληρωμάτων. Φυσικά χρειάζεται να υπάρχει αυτό το για καιρό κρίσης και επομένως πρέπει να έχουν ενία προσόντα τα, τα μέλη του προσωπικού και είναι απαραίτητο επίσης να έχουμε κοινέ ασκήσεις για να μπορούμε στη συνέχεια να δουλεύουμε σε θέατρα ε, επιχειρήσεων. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι από τον καιρό η ειρήνης. Αυτό γίνεται φυσικά με εθνικό τρόπο. Η, η εκπαίδευση των ε, του υπταμένου προσωπικού είναι κάτι που γίνεται σε εθνικό επίπεδο, αλλά εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε ένα με ενιαίο τρόπο σε εν καιρό ειρήνης. Αυτά λοιπόν και αν έχετε περισσότερα ερωτήματα για το πρώτο αυτό στοιχείο θα επανέλθουμε στις ερωτήσεις. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να πω για την ιέτηση e είναι ότι υπάρχουν θετικά αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από την δράση του μου. E με το να συνεργάζεστε σε καθημερινό επίπεδο, βλέπετε τι κάνουν και οι άλλοι και μπορείτε να φτιάξετε περισσότερη εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της ομάδος. Βλέπουμε ότι αυτό δεν είναι κάτι που είναι απλώς γραπτό στα εγχειρίδια, είναι κάτι το οποίο γίνεται στην πραγματικότητα. Υπάρχει μια αλληλεγγύη η οποία δημιουργείται. Γιατί εργαζόμαστε πράγματι, όπως είπα, σε, σε επίπεδο συνεργασία καθημερινά. Μπορούμε να το δούμε αυτό και σε καιρό ειρήνης. Γιατί όταν υπάρχει η ανάγκη να μεταφέρουμε, παραδείγματος χάρη, προσωπικό στο Αφγανιστάν ή στην Αφρική και χρειάζονται αεροσκάφη, όλοι οι άλλοι εταίροι κάνουν ό,τι μπορούν για να τους δώσουν τα αεροσκάφη αυτά. και σε ε, περίοδο κρίσης είχαμε εμπλακεί στις επιχειρήσεις στη Λιβύη, υποστήριξη στην ε, επιχείρηση αυτή και εφέτος και πέρσι στην επιχείρηση Σέρβαλ στο Μαλί. Και φυσικά η ATC συμμετέσχε με τα διαθέσιμα της μέσα το που είναι σημαντικό να κατανοήσετε είναι ότι κάποια κράτη συμμετέχαν, συμμετέσχαν λιγότερο στην υποστήριξη αυτών των επιχειρήσεων από τα άλλα. Αυτό είναι φυσιολογικό. Αυτό δεν εμπόδισε όμως τα κράτη αυτά στο να σταθούν αρρωγή στα κράτη-μέλη που εμπλάξαν περισσότερο στις επιχειρήσεις αυτές. Αυτό ήταν μια έκφραση αλληλεγγύης. Και έτσι δουλεύουμε. Και επιπλέον Έχω το παράδειγμα της Γερμανίας, στην Αφρική, που έδωσαν στη Γαλλία, που ήταν η επικεφαλής ομα, ε, χώρα στο Σερβάλ, δώσανε αεροσκάφη, Airbus, χωρίς να ζητήσουν να υπομειστεί η Γαλλία το κόστος. Αυτό το έκαναν σαν μια πράξη αλληλεγγύης. Μπορεί να σας φαίνεται μια αντιμερή συμφωνία, αλλά επειδή συνεργαζόμαστε κάθε μέρα με τη Γερμανία, στον τομέα αυτό ε, της, ε, των αερομεταφορών και του ανεφοδιασμού αεροσκαφών στον αέρα, επειδή το κάνουμε αυτό σε καθημερινό επίπεδο, ήταν έτοιμοι να κάνουν αυτή τη συγκεκριμένη γενναιόδορη προσφορά. Αν προχωρήσουμε λίγο περισσότερο, Θέλω να τονίσω ότι εμείς συμμετέχουμε σε καθημερινό επίπεδο στην ανάπτυξη της ε, Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας. Έχουμε σε στόχο να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν κοινοί κανόνες για τις ε, αερομεταφορές. Σας έδωσα το παράδειγμα των αδειών υπέρπτυσης που είναι χαρακτηριστικό γιατί έτσι μπορούμε να επεκτείνουμε μια τέτοια ιδέα, όπως έκανε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας, που το επεξέτεινε και στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα προχωρούμε σε μια κοινή συμφωνία μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ε, άδειε αυτές. Δεύτερο στοιχείο, ε, <clears throat> είμαστε πλήρως εμπλεκόμενοι στην αξιοποίηση του Α400M, του μεγάλου μεταγωγικού αεροσκάφους και επίσης θέλουμε να αναπτύξουμε την ε, ανάπτυξη μιας ικανότητας εναέριου ανεφοδιασμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και φυσικά υπάρχει και η πτυχή της ε, κατάρτισης που μπορούμε να κάνουμε για τα θέματα της ε, ΕΠΑ. Λοιπόν, να σας πω πού ακριβώς βρισκόμαστε, τι ακριβώς κάνουμε. Ονομαζόμαστε Ευρωπαϊκό Επιτελείο Ενερίων Μεταφορών. Ουσιαστικά είμαστε κράτη-μέλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον ΝΑΤΟ που θελός κάποια στιγμή αποφασίσαμε να συνεργαστούμε στενά για το pooling and sharing, τη συνεκμετάλλευση και την κοινή χρήση δυνατοτήτων κυρίως στους τομείς των αεροπορικών μεταφορών και του ενέργειου ανεφοδιασμού καυσίμων. Συνεργαζόμαστε όμως προφανώς όπως βλέπετε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, με το ΝΑΤΟ, με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Συντονισμού Κινήσεων, με τον Ευρωπαϊκό Στόλο Εναέρων Μεταφορών. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή να δημιουργήσουμε άλλο επικάλυψη αρμοδιοτήτων, αλλά να εργαστούμε πιο έντονα και να συνεργαστούμε μάλλον από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τώρα τη βάση μας στο Εντόβεν, αν διατηρήσουμε τους αριθμούς που έχουμε αυτή τη στιγμή, θα είμαστε σε θέση στο μέλλον να χρησιμοποιήσουμε 100 Α400M αεροσκάφη μας έχουν, δει συγκεκριμένες, μας έχουν δοθεί συγκεκριμένες αρμοδιότητες όσον αφορά το pooling and sharing προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα όσον αφορά τα αεροσκάφη αυτά pooling and sharing όσον αφορά τον εξοπλισμό των αεροσκαφών αυτών, κοινή κατάρτιση όσον αφορά τα πληρώματα και τους επόμενους μήνες θα χρησιμοποιήσουμε τα πρώτα A400M από τη βάση που έχουμε στη Γαλλία. Θέλουμε στα πλαίσια του ATC να χρησιμοποιήσουμε τις νέες αυτές δυνατότητες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε τόσο τα αεροσκάφη αυτά, Α400M, αλλά και τα πετρελοφόρα αεροσκάφη πολλαπλού σκοπού, MRTT, τα οποία κατασκευάζονται στην Ισπανία, και θα καταφέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο να διευκολύνουμε τη δράση μας και να γίνουμε κάπως πιο αποτελεσματικοί. Βέβαια θα πρέπει να έχουμε το ύψιστο δυνατό επαγγελματικό επίπεδο όσον αφορά τόσο τις αεροπορικές μεταφορές και όσον αφορά τον ενέριο ανεφοδιασμό καυσίμων. Τώρα, όσον αφορά την εκπαίδευση, βασιζόμαστε πάλι εδώ πέρα σε κάποιες πρωτοβουλίες που έχουμε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούμαστε στην Ισπανία, αλλά θα πάμε και στη Βουλγαρία το καλοκαίρι. Προσπαθούμε να καταρτήσουμε προσωπικό. Στο 2012 είχαμε έξι συμμετέχουσες χώρες, 8 το 2013 και 10 το 2014. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο εγχείρημα έχει στεφθεί με επιτυχία και βλέπουμε ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες χώρες οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα EATT, σε αυτό το ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Και αυτό γιατί συνειδητοποιούν όλα τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν ότι προφανώ του συμφέρει και από οικονομική πλευρά να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο κοινό πρόγραμμα εκπαίδευση. Βλέπετε εδώ πέρα και κάποια άλλα αριθμητικά δεδομένα όσον αφορά το EAATTC, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εχμή, ε, όσον αφορά στην κατάρτιση τακτικών αερομεταφορών. Μέσω όλων αυτών των πρωτοβουλειών σε μειωμένη κλίμακα πέντε κράτη-μέλη ε, επί του παρόντος 7 στο μέλλον, μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουμε κάποιους ε, κανόνες και κάποιες μορφές συνεργασίας που θα αποφελήσουν πολλά περισσότερα κράτη-μέλη στο μέλλον. Όσον αφορά δηλαδή αυτούς τους καονισμούς απασχόλησης, όσον αφορά τις μεθόδους ε, κατάρτισης και το καθεξής. Θα υπάρχουν στο μέλλον όλο και περισσότερα κράτη-μέλη που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προγράμματα αυτά, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα μπορούμε να συνεργαζόμαστε από στρατηγικής πλευράς πολύ καλύτερα και όλο και περισσότεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα τώρα να εκφράσω και τις δικές μου προσωπικές απόψεις για τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας όσον αφορά την πρωτοβουλία Pooling and Sharing, συνένωσης και κοινή χρήσης στα πλαίσια, του EATC. Τα πράγματα νομίζω ότι είναι πολύ απλά, δυστυχώς δεν φαίνονται πολύ καλά στη διαφάνεια, Στα πλαίσια του pooling and sharing και οποιασδήποτε τέτοιες πρωτοβουλίες χρειάζεται καταρχάς μια έντονη πολιτική βούληση από δύο τουλάχιστον χώρες. Δεν μπορεί κανείς να συνεργαστεί με τον εαυτό του ή ακόμα και γινόταν κάτι τέτοιο θα ήταν ιδιαίτερα περιορισμένο. Πρέπει να συνεργαζόμαστε με κάποιον άλλον εταίρο. Καταρχάς λοιπόν μια πολύ σημαντική έντονη πολιτική βούληση. Δεύτερον, χρειάζεται κανείς μία σαφή έννοια, ένα σαφή ορισμό όσον αφορά το ζήτημα των στρατιωτικών δυνατοτήτων, δηλαδή ποιο είναι το πλαίσιο εκείνο για να καταφέρουμε να έχουμε ένα αποτελεσματικό pooling and sharing. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κενό πλαίσιο, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια δομή η οποία σε καθημερινή βάση να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν. Έτσι λοιπόν Βλέπετε ότι στα πλαίσια του ATC, στα πλαίσια της δημιουργίας του ATC, είχαμε δύο πυλώνες, τον επιχειρησιακό πυλώνα και τον λειτουργικό πυλώνα. Ξέρω ότι η διάρθρωση αυτή, η δομή αυτή μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη. Τρίτον, κάτι το οποίο ανέφερε και ο πρόεδρος Ντανζό, αν πραγματικά θέλετε τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν στον τομέα των στρατιωτικών δυνατοτήτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουν αυτά τα κράτη από τη μια ότι πρέπει να εκχωρήσουν κάποιες αρμοδιότητες και από την άλλη θα πρέπει να γνωρίζουν πρώτον ότι προοδευτικά θα πρέπει να δεσμευτούν όλο και περισσότερο για την πρωτοβουλία αυτή, δηλαδή δεν χρειάζεται να εκχωρήσουν τα μέσα του στρωτικά αμέσω, αλλά προοδευτικά σταδιακά μπορούν να εκχωρούν τα μέσα αυτά και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν δεύτερον ότι όλη η δικασία είναι και αναστρέψιμη. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή ένα κράτος μέλος εκχωρεί αεροσκάφη στα πλαίσια του EATC, ανά πάσα στιγμή μπορεί να μας πει ότι από τα αεροσκάφη τα οποία έχει εκχωρήσει χρειάζεται να πάρει πίσω δύο αεροσκάφη για κάποια εθνική αποστολή. Δεν χρειάζεται καν να δικαιολογήσουν την απόφαση αυτή ανάκληση των αεροσκαφών. Πρέπει απλώ να στείλουν ένα email και να μα λένε ότι, για παράδειγμα, αύριο θα χρειαστεί να ανακαλέσουμε δύο από τα αεροσκάφη που σα έχουμε δώσει γιατί τα χρειαζόμαστε για κάποιου εθνικού λόγου. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μία προοδευτική εκχώρηση αρμοδιοτήτων και μέσων, η οποία, όπω σα είπα, είναι αστρέψιμη. Το τίμημα, βέβαια, στην περίπτωση αυτή, είναι ότι θα πρέπει να εκχωρηθεί και μια κάποια αρμοδιότητά του προ την κεντρική αυτή δομή. Ένα ακόμα σημείο, το οποίο ενδεχομένω να είναι ευνόητο, αλλά θεωρώ ότι είναι θεμελιώδου σημασία. Είναι μια μάχη που δίνουμε σε καθημερινό επίπεδο. Αν πραγματικά θέλετε μια τέτοια δομή με στρατιωτικά μέσα να είναι όντω αποτελεσματική, θα πρέπει η διάρθρωση αυτή, η δομή αυτή, το επιτελείο αυτό, η διοίκηση να μπορεί να ενσωματωθεί στα πλαίσια της αλυσίδας διοικητικής μέρημνας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Στα πλαίσια του EATC, στην περίπτωση μάλλον του EATC, εμείς δίνουμε κάποιες συγκεκριμένε διαταγές ως προς τις επιμέρους μονάδες μας, Υπάρχει όμως ένα γενικότερο πλαίσιο και γίνεται αποδεκτό κατά αυτόν τον τρόπο από ένα κράτος μέλος ότι οι εθνικές στρατιωτικές τους δομές μπορούν να λάβουν πλέον εντολές από ένα κεντρικό επίπεδο προκειμένου από το Eindhoven. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου να έχουμε μια αποτελεσματική στρατιωτική συνεργασία. Το τελευταίο σημείο το οποίο θέλω να θίξω είναι ότι, και αυτό μπορεί να σας φανεί τεχνικό, αλλά χρειαζόμαστε να χρησιμοποιούμε ένα κοινό πλαίσιο πληροφορικής. Ξέρετε πώς λειτουργούν τα πράγματα αυτά, δεν μπορούμε να αποφύγουμε σε καμία περίπτωση την πληροφορική. Πέρα από τα εθνικά συστήματα πληροφορικής θα πρέπει να επιτρέψετε τη λειτουργία ενός κοινού μέσου πληροφορικής προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση και κοινή συνεργασία των δυνατοτήτων. Και κάτι ακόμα, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, το βλέπετε εδώ πέρα με αυτό το θετικό πρόσημο, στη διαφάνεια. Κάθε φορά που μιλάμε για pooling and sharing στρατιωτικών μέσων ή δυνατοτήτων, αυτή μπορεί πραγματικά να είναι αποτελεσματική μόνο αν η επικεφαλή των ενόπλων δυνάμεων για οποιοδήποτε σώμα, ναυτικό ή πολεμική αεροπορία συμμετέχει, αν συμφωνούν οι άνθρωποι αυτοί να συνεργαστούν, γιατί διαφορετικά η συνεργασία αυτή δεν θα είναι σε καμία περίπτωση αποτελεσματική. Πρέπει να εμπλέκονται, να μπορούν να συμμετέχουν και οι αρχηγοί των διαφόρων στρατιωτικών επιτελείων. Αυτό το βλέπουμε και με την Ισπανία, για παράδειγμα. Ε, ο επικεφαλής της πολεμικής αεροπορίας της ε, Ισπανίας συνέβαλε πάρα πολύ καθοριστικά στην ε, συμμετοχή της χώρας του στο EATC. Ο πτέραρχος Ανάης συμμετέχει λοιπόν άμεσα και είναι πάρα πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, να μπορούμε να έχουμε τους επικεφαλείς ενόπλων δυνάμεων κάθε χώρας ε, να επιθυμούν ουσιαστικά αυτοί να συμμετέχουν στο EATC. Προτού ολοκληρώσω να σας πω το ακόλουθο. Προφανώς παραμένουν ακόμα πολλές προκλήσεις. Δεν θα επιστέλθω σε πολλές λεπτομέρειες. Πάντως ε, δημιουργήθηκε το EATC πριν από 3-3,5 χρόνια. Ξεκινήσαμε από το 0. Και βέβαια πρέπει να παγιώσουμε σιγά σιγά τις διαδικασίες μας, να καταφέρουμε να βελτιώσουμε την ολοκλήρωση των συμμετεχόντων κρατών μελών και θα πρέπει να πείσουμε τελικά τους εμπλεκουμένους να συμμετέχουν περισσότερο και να επενδύουν περισσότερο στο EATC και να επιθυμούν να συνεργαστούν όλο και περισσότερο μαζί μας. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, Αναφέρθηκα στην προσχώρηση της Ισπανίας και της Ιταλίας, θεωρητικά είναι εύκολη, αλλά καταλαβαίνετε ότι στην πράξη θα πρέπει να συνοδεύσουμε τα κράτη αυτά και θα πρέπει τελικά να δέσει μαγιονέζα, να μου το επιτρέπετε. Δηλαδή, το αποτέλεσμα τελικών είναι θετικό για όλους. Ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε εδώ πέρα για την συμμετοχή και τη συνεργασία πολλών κρατών, οι οποίοι εκχωρούν ουσιαστικά τις δικές τους αρμοδιότητες, επενδύουν μέσω προσωπικού, μέσω μέσων, μέσω αλλαγών και τροποποιήσεων που αναγκαστικά κάνουν στις διαδικασίες τους. Αυτό είναι δαπανηρό από πολλές πλευρές, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θέλουν να δούνε απτά αποτελέσματα. Με τη συμμετοχή λοιπόν της Ισπανίας και της Ιταλίας θέλουμε και να εξασφαλίσουμε ότι θα υποφεληθεί το EATC, αλλά θέλουμε να αποφελούνται και τα επιμέρους μέλη του οργανισμού αυτού. Αυτή είναι η συνεχής πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε. Ένα τελευταίο τώρα σημείο, ένα μήνυμα το οποίο θέλω να σας στείλω, όσον αφορά το πόσο ελκυστικός μπορεί να είναι αυτός ο οργανισμός, δημιουργώντας ένα πολυεθνικό τέτοιο όργανο στις κάτω χώρες ή οπουδήποτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να προσελκύσουμε προσωπικό ανθρώπους οι οποίοι θα επιθυμήσουν να έρθουν με τις οικογένειές τους, να κατασταθούν στο Eindhoven και να εργαστούν για μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και το ζήτημα των σχολείων είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Υπάρχουν ε, πολλές οικογένειες οι οποίες ναι μεν θέλουν να έρθουν στο Eindhoven, αλλά θέλουν να πάνε και τα παιδιά τους στα καλύτερα δυνατά σχολεία, θέλουν να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση στα παιδιά αυτά σε πολλές και διάφορες γλώσσες, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι χρειαζόμαστε και ευρωπαϊκά σχολεία. Στην περίπτωση του EATC τι έχουμε, έχουμε το Ευρωπαϊκό Σχολείο του ΜΟΛ στο Βέλγιο, το οποίο ανταποκρίνεται πολύ καλά στις ανάγκες μας. Δεν βρισκόμαστε όμως εδώ στη σωστή κατηγορία. Εμεί θέλουμε να κάνουμε αιτήσει προς την ε, κατηγορία παριθμών 1, δηλαδή διδασκαλία να διασφαλίζεται στη μητρική γλώσσα και δεν θέλουμε τα δίδακτρα να καταβάλλονται από τις οικογένειες. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη λεγόμενη κατηγορία παριθμών 3. Εμείς θα υποβάλουμε εκ νέου μία αίτηση προκειμένου να καταφέρουμε να αναβαθμιστούμε στην κατηγορία 1. Ολοκληρώνω λοιπόν σε αυτό το σημείο. Ελπίζω και εύχομαι να γνωρίζετε πλέον καλύτερα ποιοι είμαστε, τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Πάντως, εν δυνάμει μπορούμε να υποσχεθούμε πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο για την προσχώρηση των νέων κρατών μελών και την δυνατότητα χρησιμοποίησης νέων μέσων, αλλά μπορούμε να προωθήσουμε όλο περισσότερο την κοινή πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας. Και όσον αφορά την δήλωση της 20ης Δεκεμβρίου του Συμβουλίου, όντως συμφωνούμε και εμείς ότι θα μπορούσε η μέθο αυτή να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες στρατοτικές δυνατότητες και σε άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα στον τομέα της θάλασσας ή στην επιτήρηση όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές, νομίζω ότι το δικό μας το μοντέλο θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλες πρωτοβουλίε Και να επαναλάβω και κάτι ακόμα, αποτελεί και πάλι αυτό προσωπική άποψη, εργάζομαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια στα πλαίσια του ε, στρατού, της πολεμικής αεροπορίας. Έχω δει τελευταία 30-40 χρόνια πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Σήμερα περισσότερο από ποτέ σας το λέω ότι η συνεργασία δεν αποτελεί πλέον απλώς επιλογή. Είναι μια πραγματική ανάγκη και Ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Επιτελείο Νερίου Μεταφόρων μπορεί να αποτελέσει ένα θετικό παράδειγμα για αυτή τη μελλοντική συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Ήταν εξαιρετικά σαφή, συγκεκριμένη, πληρέστατη παρουσίασή σας. Έχω μια ερώτηση. Αυτονόητο φαντάζομαι είναι ότι τα κράτη είναι αυτά που σας ε, δίνουν εντολή, σας αναθέτουν καθήκοντα στο πλαίσιο του συλλογικού σχεδιασμού, σε ποιο σημείο ε, έρχονται σε εσά. Μιλάω για τις σχέσεις ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης ή νατοικές ε, ή ευρωπαϊκές δομές. Πότε στρέφονται σε εσάς. εφόσον είστε ένα σημαντικό κρίκο όλων των επιχειρήσεων, το βλέπουμε και στι ε, συζητήσει, ιδίω για την κεντροαφρικανική δημοκρατία, για το ενδεχόμενο ευρωπαϊκή επέμβαση. Υπάρχουν σημαντικέ δυσκολίε στον τομέα τη επιμελητία. Πρώτον, απευθύνεται κανεί απευθεία σε εσά, από κάποιο συλλογικό όργανο, από αυτού του οργανισμού νατοικού ευρωπαϊκού και αν ναι, σε ποια χρονική στιγμή ή αποκλειστικά τα κρατημέλη είναι αυτά τα οποία πολύ νωρίς τελικά, ε, μάλλον πολύ μετά σε ύστερο στάδιο, έρχονται σε επαφή μαζί σας, αφού δηλαδή έχει εγκριθεί παραδείγματο χάρη στρατηγική για την Κεντρία Αφρικανική Δημοκρατία. Αυτό είναι το δικό μου ερώτημα. Θα ακούσουμε και τους άλλους ε, βουλευτές και θα σας δώσουμε το λόγο για να απαντήσετε. Ο κύριος Uh, thanks for presentation. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Η ε, γενική άποψη είναι ότι όλη η καλή δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ε, το χθες. Το θέμα που μας απασχολεί σήμερα είναι είναι έτοιμη να πολεμήσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Και αν υπάρχει θέληση να πολεμήσει κανείς, τότε πρέπει να έχουμε υπόψη μας το αύριο. Και όχι μόνο την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύξει, να αναρμονίσει το οτιδήποτε, αλλά την ικανότητά της να αναλάβει δράση. Γιατί μόνο αυτό ε, μετράει, παραδείγματο χάρη, σήμερα στη Μόσχα. Μόνο αυτό, αν είμαστε σε θέση να δράσουμε. Οι διεθνείς πολιτικές ασφάλειας δεν ορίζονται από τα χαρτιά, αλλά από τη δράση και δεν είναι του χθε, αλλά πρέπει να είναι του σήμερα και του αύριο. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Κύριε Βανόρντεν, είδα να σχηματίζετε ένα μηδία με ικανοποίηση στα χείλη σα. Φαντάζομαι ότι αυτά που ακούσατε, δηλαδή το συνδυασμό ρεαλισμού και υπάρχει και έκφραση εγώ want my planes back, θέλω πίσω τα αεροπλάνα μου. Θα σας αρέσουν όλα αυτά, είμαι σίγουρος. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και τον υποπτέραρχο για την πολύ ξεκάθαρη εξήγηση. Πρέπει να σας πω ότι πραγματικά και είμαι υπέρ των εφιών αποδοτικών, οικονομικών, συνεργατικών πρωτοβουλειών. Υπάρχει μακρά ιστορία τέτοιων πρωτοβουλειών ε, για την υποστήριξη του ΝΑΤΟ επί πολλές δεκαετίες και αυτή είναι μια ακόμη τέτοια πρωτοβουλία. Θέλω να πω όμως εφές εξ αρχής ότι το πρόβλημα είναι ότι όταν μπει η λέξη ευρωπαϊκός πάνω από κάτι, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να το καπελώσει κατά κάποιο τρόπο, σαν να είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ βρήκα πάρα πολύ ωραία την παρουσία σας μέχρι τις δυο τρει τελευταίες σας φράσεις ε, είπατε ότι μπορεί να βοηθήσει βέβαια, ε, να προωθηθεί και η ΕΠΑ, η κοινή πολιτική μάλλον ασφάλειας και άμεσης. Ξέρετε, η κρίση στην Ουκρανία υπογράμμισε την ανάγκη για το ΝΑΤΟ, για ένα αναζωογονημένο ΝΑΤΟ με ενή άποψη. Και δεν θέλουμε να αποσπαστεί προσοχή μας με αυτή την ανόητη ιδέα ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρεμβαίνει αμυντικά κάπου στον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ χρήσιμη μπορεί να είναι με τα μη στρατιωτικά τη μέσα και πολλές άλλες πτυχές, διαχείριση κρίσεων κτλ. Όχι όμως να αναμειχθεί στην άμυνα, στα αμυντικά ζητήματα. Οτιδήποτε ενθαρρύνει λοιπόν κάτι τέτοιο, φοβούμαι ότι με βρίσκει αντίθετο και ανησυχώ πάρα πολύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια ταυτότητα, ε, μάλλον μια κρίση ταυτότητα ε, και προσπαθεί ε, να εξελιχθεί σε ένα είδος κρατικής οντότητας. Η δική σας πρωτοβουλία, ο δικός σας οργανισμός είναι διακυβερνητικός. Το είπατε και το καταστήσατε απόλυτα σαφές. και μπορεί οποιοδήποτε άλλο οργανισμό να εμπλουτίσει, ε, μάλλον να χρησιμοποιήσει τα μέσα του. Θα ήταν λάθος να πούμε ότι είναι ευρωπαϊκού τύπου ε, οργανισμός, γιατί δεν είναι. Έχω ένα-δύο ερωτήματα. Θα μπορούσατε να διευκρινίσετε τη σχέση μεταξύ EATC και του Κέντρου Συντονισμού Κίνησης στο Αιτχόφεν. Νομίζω 25 είναι οι συμβαλόμενοι και είπα μεταξύ αυτών. Ενδιαφέρον, κάτι, ενδιαφέρον αυτό και δεν ξέρω αυτά τα δύο κέντρα πώς ε, συνδέονται αν συνδέονται. Επίσης μιλήσατε για την τυποποίηση των διαδικασιών. Δεν βοηθά το ανατοϊκό πρότυπο εδώ. Γιατί να επανεφεύρουμε συνεχώς τον τροχό στα θέματα της διαλειτουργικότητας και της τυποποίησης. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κάποια πρότυπα. Και σε ό,τι αφορά το διεθνές καθεστώς, Αναφερθήκατε σε διάφορους τομείς ε, που πολύ χρήσιμη ήταν η συνεισφορά του η ATC, η γαλλική επιχείρηση στο Σαχέλ, οι γαλλικές επιχειρήσεις θα έλεγα στο Σαχέλ. Ξέρετε και επειδή και το Ηνωμένο Βασίλειο βοήθησε με προσφορά μέσων πόρων, γιατί να μην βασιστούμε απλά στο EATC και θα πρέπει να περνάμε, ε, να πηγαίνουμε πιο πέρα για την απαιτούμενη περαιτέρω ε, κινητοποίηση που ζητούν οι γαλλικές δυνάμεις. Στρατηγία μου. Είναι πολλά τα ερωτήματα <clears throat> που τέθηκαν. Το τελευταίο ερώτημα θα αντιμετωπίσω πρώτα, αν μου επιτρέπετε, για την ε, επιχείρηση Σερβάτ στο Σαχέλ. Έχετε δίκιο σε ό,τι αφορά την υποστήριξη σε ό,τι της επιχείρησης στο Σαχέλ, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι τέτοιου είδους επιχειρήσεις βρίσκονται ουσιαστικά στο ανώτατο όριο της ε, ακτίνος δράσης της EATC. Μιλάτε για χιλιόμετρα, <clears throat> για ε, χιλιάδες χιλιόμετρα μετα, με, μακριά από την Ευρώπη και μεταφορά στρατευμάτων. Για την προετοιμασία της επιχείρησης Serval ...75 με 80% της αερομεταφοράς έγινε με ναύλωση αεροσκαφών. Τα μεγάλα Αντόνοφ ήταν τα μόνα αεροσκάφη που ήταν σε θέση να μεταφέρουν τόσου πόρους στο Σαχέλ. Στη συνέχεια υπήρχε ένα αριθμό από συμμάχου όπω είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδά και οι, το, οι Ηνωμένες Πολιτείες με τα e ΕΣΥ 17 που έδωσαν το υπόλοιπο 10-15% της ε, ανάγκης αερομεταφοράς και 5% δόθηκε από την EATC. Και όχι γιατί οι χώρες μας, η Γαλλία, η Γερμανία κτλ. δεν θέλαν την EATC, γιατί δεν παίρνονται σε λεπτομέρειες, αλλά το προφίλ των αεροσκαφών που έχουμε για ε, μεταφορές βαρέων φορτίων σε μεγάλη ακτίνα δράση, αυτό δεν είναι κάτι που έχουν πια τα κράτη-μέλη του e ATC. Δεν έχουμε τέτοια αεροσκάφη. Επομένως η Γαλλία χρησιμοποίησε τα μέσα τα οποία θεώρησε ότι να χρησιμοποιήσει, απευθύνθηκε σε εξωτερικούς παρόχους που είχαν μεγαλύτερα αεροσκάφη. Για το γενικό σας τώρα ερώτημα. Η σύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και του EATC. Κατανοείται φυσικά ότι δεν μπορώ εγώ να πάρω μια πολιτική θέση για τα θέματα αυτά. Αλλά από τεχνική άποψη αυτό το οποίο μπορώ να πω και για να απαντήσω και στο ερώτημα του Πρόεδρου Ντονζόν μέχρι στιγμής δεν μας έχει ζητήσει κανείς ούτε το ΝΑΤΟ ούτε η, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιος να σχεδιάσουμε την υποστήριξη μιας επιχείρησης. Δεν έχει γίνει ακόμα. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι κάποια κράτη-μέλη ζητούν από την EATC να σχεδιάσει υποστήριξη μιας επιχείρησης. Επομένως προετοιμάζετε αεροσκάφη, ότι προσπαθείτε να έχετε ώστε να τον περισσότερα μέλη να βοηθήσουν για τη μεταφορά στρατευμάτων, χάρη στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία κτλ. Εμείς λοιπόν εμπλεκόμαστε μέσω των κρατών μελών που ανήκουν στην EATC. Δεν ζητάει κανείς κατευθείαν από εμά να κάνουμε κάτι. Και σε ό,τι αφορά τη συνολική αντίληψη και το νομικό πλαίσιο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιος σαφής μηχανισμός βάσει του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε κατευθείαν να ζητήσει τη βοήθεια του EATC. Και αν συνέβαινε κάτι τέτοιο βέβαια, θα έπρεπε να περάσουν από τα λεγόμενα κράτη χορηγούς του EATC, Γαλλία, Γερμανία και τα λοιπά και τότε το κράτος αυτό <clears throat> θα μπορούσε να αναλάβει την αντιμετώπιση αυτής της αίτησης μεταφορών. Αυτά λοιπόν για να σας πω δεν είναι ότι δεν υπάρχει τέληση. Και ουσιαστικά ε, υπάρχει η αίτηση μόνο για 2,5 χρόνια. Δεν μας έχει ζητήσει κανείς να συμβάλλουμε σε μια υποστήριξη επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα με την επιχείρηση για την κεντροαφρικανική δημοκρατία όπου μπορεί να υπάρξει μια άμεση αίτηση για το, ε, η αίτηση να συμβάλλει στο συντονισμό των αερομεταφορών σε αυτή την επιχείρηση. Και δεν είμαι εδώ για να σας πω ότι θα συμβάλλουμε ή δεν θα συμβάλλουμε, αλλά δεν θέλω να σας δώσω την εντύπωση αλαζονίας. Αυτό που κάνουμε στο δικό μας επίπεδο, τα πέντε κράτη και αύριο τα εφτά κράτη, στον τομέα μας ε, αρμοδιότητας, είναι να διαρθρώνουμε σωστά τις ικανότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό πιστεύω ότι μπορεί να συμβάλλει σε μια διαδικασία εκ των κάτω προς τα άνω στην διαμόρφωση μιας συνολικής ικανότητας για όλη την Ευρώπη. Αλλά δεν θέλουμε εμείς να συγκεντρώσουμε τα πάντα στο Eindhoven. Θέσατε ένα ερώτημα για το κέντρο συντονισμού των μετακινήσεων των μεταφορών στην Ευρώπη και οι δύο, είμαστε στο Eindhoven. Και είναι μεγαλύτερος αυτός ο φορέας, καλύπτει 25 ε, χώρες είμαστε πέντε. Η μεγάλη διαφορά βρίσκεται στο ότι το MCC, το Κέντρο Μεταφορών στην Ευρώπη, αντιμετωπίζουν όχι μονάχα εναέριες μεταφορές, αλλά και χερσαίες μεταφορές και θαλάσσιες μεταφορές. Επομένως υπάρχει συνεργασία στο pooling και sharing και για θαλάσσιους πόρους. Κάνουν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την ε, μετακίνηση δυνάμεων από το Αφγανιστάν στο αεροπορικό επίπεδο είναι διαφορετική η δράση μας από το MCC, γιατί το MCC είναι κατά κάποιο τρόπο ένας διαμεσολαβητής. Έχουν προσφορές από τη μία μεριά που έρχονται από τα κράτη-μέλη. Λέει κάποιος έχω ένα ελεύθερο φορτηγό, ένα άδειο φορτηγό πλοίο ή ένα άδειο φορτηγό αεροπλάνο και από την άλλη μεριά υπάρχουν αυτοί οι οποίοι ζητούν πόρους μεταφορών. Δεν κάνει όμως τίποτα περισσότερο. Ενώ η ETC εμείς συνεργαζόμαστε από την αρχή, από την φάση σχεδιασμού μιας αποστολής. Υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός λοιπόν συνεργασίας και ολοκλήρωσης πολύ πιο ισχυρό στη δική μας περίπτωση γιατί ο στόχος δεν είναι ακριβώς ο ίδιος, ο στόχος είναι να μπορούμε να εκτελούμε αποστολές ημέν για τους δε και είναι πολύ πιο έντονη αυτή η συνεργασία. Το MCC βέβαια κάνει πολλά πράγματα, βοηθάει, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και για την τυποποίηση που αναφέρθηκατε. Ίσως ήμουν κάπως παραπλανητικός. Θα πρέπει να λέω εναρμόνιση διαδικασιών γιατί τα STAN acts, οι πράξεις τυποποίησης του ΝΑΤΟ εξακολουθούν να ισχύουν. Είμαστε όλοι μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά υπάρχουν τομείς όπου δεν επαρκείς η stan acts όπως λέγονται όπως παραδείγματος χάρη για τη χρήση αλεξιπτωριστών. Έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να στείλουμε Γερμανούς, να ρίξουμε ε, Γερμανούς αλεξιπτωριστές ε, από ένα γαλλικό σε 160 ή από ένα βελγικό σε 130 και δεν θέλω να πω σε περισσότερες λεπτομέρειες. φυσικά εμεί κατά τα άλλα ακολουθούμε το γενικό πλαίσιο του ΝΑΤΟ και των ΣΤΑΝΑΤΣ. Δεν ξέρω αν απάντησα όλα τα ερωτήματα. Ναι, και το θέμα της ε, ε, ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πολεμήσει. Μα δεν θα το απαντήσω εγώ αυτό το ερώτημα. Ως EATC πάντως, και εκεί βρίσκεται η ομορφιά του η Τα κράτη που βρίσκονται στην αίτηση έχουν διαφορετικές φιλοδοξίες μέσω της αίτηση. Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας που λέει όλοι πρέπει να κάνουν το ίδιο πράγμα. Υπάρχει ένα ευρύ πλαίσιο, αλλά ο καθένας έχει διαφορετικές φιλοδοξίες. Η δυνατότητα παρέμβαση δεν είναι ίδια για όλα τα κράτη-μέλη. Όλοι όμως συμμετέχουμε στο Αφγανιστάν. Πολλά από τα κράτη μας πηγαίνουν στην Αφρική Έτσι λειτουργεί λοιπόν το σύστημα αυτό. Εμείς κάνουμε ό,τι μας ζητάνε οι κυβερνήσει μας να κάνουμε. Αλλά υποστηρίζουμε επιχειρήσεις κάθε μέρα, κάθε νύχτα σε όλο τον κόσμο. Αναφέρθηκε το Αφγανιστάν, αναφέρθηκε το Κωσυφοπέδιο, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το Μαλί, το Νότιο Σουδάν. Κάποιοι από εμά είναι εκεί πέρα για να μπορέσουν να ε, εκενώσουν προσωπικό από τον Νότιο Σουδάν και να το φέρουν στη Γερμανία. Είμαστε λοιπόν ένα εργαλείο για μια ομάδα κρατών και προσπαθούμε να είμαστε ένα αποτελεσματικό εργαλείο. Ευχαριστώ. Μήπως μπορώ να σας θέσω ένα ερώτημα το οποίο ίσως είναι εκτός θέματος. Μήπως θα μπορούσατε να φανταστείτε χώρες που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ ή μήχο μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν εθελοντικά να συμμετάσχουν στο EATC ή ο βαθμός εναρμόνισης που απαιτείται και η ελάχιστη πολιτική συμφωνία που απαιτείται δεν το κάνει αυτό εφικτό. Πολύ καλό το ερώτημα από αυτή την πλευρά. Τίποτα δεν ε, αποτρέπει ε, ένα κράτος ε, που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, δηλαδή της Ένωσης, να προσχωρήσει σε εμά. Μπορεί να υποβάλει πολύ απλά μια αίτηση, στέλνοντας μια επιστολή στο EATC. Συνήθως ε, το στέλνει ο αρχηγός ε, της αεροπορίας, του Γενικού Τηλεαεροπορίας ή τέλος πάντων κάποιος από την αρχή, από την χώρα αυτή και λέει θέλουμε να προσχωρήσουμε και έπειτα γίνεται ε, αξιολόγηση. Δεν υπάρχει κάποιο έγγραφο που να ορίζει ότι θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκό ή όχι κράτος. Για να πάω και λίγο πιο πέρα, ίσως να ακούσατε μια ομάδα σκανδιναβικών χωρών, βόρειων χωρών που αποφάσισαν να συνεργαστούν. Νορτάφκο λέγεται αυτή η ομάδα. Σε αυτήν την ομάδα υπάρχουν και ευρωπαϊκά, μάλλον και μέλη της Ένωσης και χώρες που δεν είναι μέλη της Ένωσης. Και παραλαμβάνω, τίποτα δεν αποκλεί τον δεχόμενο να προσχωρήσουν στο EATC. Γιατί το έχουμε συζητήσει και δεν είπε κανένας ποτέ σε εμά ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι σημαντικό να έχετε υπόψη ότι ακολουθούμε μια προσέγγιση πραγματικά από κάτω προς τα πάνω. Όταν δηλαδή έρχεται ένα αίτημα στο ATC, ο γνώμονας που χρησιμοποιούμε είναι τη δυνατότητά μας, την παραγωγή μας, θα τη βελτιώσει ή θα την υπονομεύσει. Φυσικά υπάρχουν και πολιτικές παράμετροι, να υπάρχει έγκριση κτλ. Έτσι βλέπουμε όμως εμείς τα πράγματα. Και για να απαντήσω στο ερώτημά σα. Εάν ο Καναδάς, είπε παραδείγματι, ζητούσε να προσχωρήσει, θα λαμβανόταν η απόφαση στο πολιτικό επίπεδο, αλλά από τεχνική πλευράς εμείς θα εξετάζαμε τι δυνατότητε του Καναδά που έχουν πολύ καλές δυνατότητες αερομεταφοράς. Και επομένως η απάντηση θα ήταν μάλλον ναι παρά όχι. Από τη δική μας πλευρά, λέει, ότι έπρεπε να ληφθούν υπόψη πολιτικές παράμετροι. Είναι και μέλος του ΝΑΤΟ, οπότε. Πρόεδρος, άλλες παρεμβάσεις δεν υπάρχουν, επομένως ε, μένουμε σε αυτά. Ευχαριστώ πολύ τον Πτέραρχο για την επίσκεψη του εδώ και τις πολύ σαφείς εξηγήσεις που μας έδωσε. σαρπαστική προσέγγιση αυτή, πολύ συγκεκριμένη. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Και τολμώ να ελπίζω ότι όσοι, εμείς, όσοι από εμάς έχουν την τιμή να είναι στην ε, επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, η πρώτη, από τις πρώτες επισκέψεις θα είναι στο γειτονικό Αιντχόβεν. Είναι κρίμα. Είστε δίπλα μας να μην επισκεφθούμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους ε, σμιναγούς, σμινάρχους. Ευχαριστώ λοιπόν τους σμινάρχους και για τη βοήθεια που παρέχεται ιδίως σε ευρωπαϊκές επιχειρήσει.